Gerbėjai κολέγος, Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητοί ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, τιμή μου που μπορώ να προεδρεύσω την ε, απογευματινή συνεδρίαση μαζί με την ε, συνάδελφό μου της Επιτροπής Ήτρε, την κυρία Πατρίσια Τόια. προεδρεύσουμε ε, στην απογευματινή συνεδρίαση και ελπίζω ότι θα είναι καρποφόρα και πλούσια η συζήτηση αυτή. Ας αρχίσουμε με την ενεργειακή πολιτική αποδοτικής χρήσης της ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις. Πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στην πλήρη ένταξη των στόχων μας προς την κατεύθυνση Ενό ευρύτερου στόχου, δηλαδή της ολοκλήρωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, την εξασφάλιση της προμήθειας της ενεργείας για καταναλωτές και επιχειρήσεις και ταυτόχρονα με μείωση των διοξιδίων του άνθρακος. Θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς με κοινέ προσπάθειες. Εάν επιθυμείτε να θέσετε ερωτήσεις, στους προσκεκλημένους ομιλητές μετά από τις παρουσιάσεις τις οποίες θα προβούν. Σας παρακαλώ να συμπληρώσετε τα κίτρινα έντυπα που έχετε, τα οποία θα συγκεντρώσουμε και θα συντάξουμε κατάλογο των αγορητών. Ο κύριος Ταγιάννη θα καθυστερήσει για, την, ε, για να έρθει στην Επιτροπή μας περίπου 20 λεπτά. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Βέρερ τον Γενικό Διευθυντή της Business Europe, ο κύριος Μπέιρερ. Ευχαριστώ, Άτσου, όπως λέτε στα λιθανικά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τη Λιθανική Βολή καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την διοργάνωση της παρούσας συνάντησης που τη βρίσκω πολύ καλή ιδέα γιατί το θέμα είναι πολύ σημαντικό στην στιγμή αυτή που βέβαια επίκειται η επίκειται η λήψη σοβαρών αποφάσεων στις 22 Ιανουαρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά βέβαια και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου καθώς επίσης και με τις κινήσεις που κάνει και το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας καθώς και για την δυνατότητα που μας δίνεται να αναπτύξουμε τις απόψεις μας διότι γνωρίζετε ότι για όλη την ε, συζήτηση περί ενέργειας είναι πολύ υψηλά τα διακυβεύματα και για τις επιχειρήσεις και για τους εργοδότες στην Ένωση. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά και υπάρχει και ένας αριθμός προβλημάτων που προκαλούνται από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε αντιμετωπίσει την υπόθεση ως τώρα. Θα χρειαστεί να αναδιοργανώσουμε τις πολιτικές, διότι δεν θα είμαστε σε θέση να εμφυσίσουμε νέα βιομηχανική πνοή στην Ήπειρο, χωρίς σημαντικές αλλαγές στην ελληνική πολιτική. Και υπάρχουν και όπως είπα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και πρώτο και προφανές βεβαίως, αλλά πρέπει να το τονίσω, είναι οι υψηλές τιμές της ενέργειας. Γνωρίζουμε ότι το φυσικό αέριο, δηλαδή οι τιμές του αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν αυξηθεί σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε ωστόσο ταυτόχρονα δει σε ανταγωνιστικές αγορές να έχουν πέσει τιμές για ηλεκτρικό ρεύμα, για παράδειγμα 37% στις χώρες του ΩΣΑ μεταξύ 2007 και 2012 ενώ έχουν πέσει κατά 4% στην, ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα φτάνουν στα 41% που, η διαφορά δηλαδή, που σημαίνει πολλές δυσχερίες για πολλές βιομηχανίες παρόμοια κατάσταση για διάφορους λόγους πάλι και στις τιμές του φυσικού αερίου. Και ε, είναι παρόμοια εικόνα και εκεί. Και αν μιλήσετε με διευθυντές βιομηχανικών εταιριών, και εγώ το κάνω πολύ αυτό, ο λόγος που δεν επενδύουν στην Ευρώπη, ένας από τους λόγους είναι οι υψηλές ε, τιμές της ενέργειας, το κόστος της ενέργειας. Βεβαίως η εικόνα είναι περιπλοκότερη, αλλά δύο τονίζουν ιδιαίτερα. υψηλέ τιμέ ενέργειας και δυσκολία πρόσβαση σε χρηματοδότηση αναλόγω τη αγορά. Έτσι λοιπόν εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των υψηλών τιμών ενέργειας. Έχουμε και επικαλυπτόμενους στόχους για την προστασία του κλίματος και άλλους περιβαλλοντικούς στόχους που ωστόσο προκαλούν στρέβλωση των μηνυμάτων που δίνουμε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και έχουμε διεξαγάγει ήδη τη συζήτηση αυτή. Βέβαια είναι χαμηλότερη η τιμή για την Ευρώπη του διευθυντήτου του αλλά αυτός είναι, ο ένας είναι ο λόγος η οικονομική κρίση και άλλοι λόγοι είναι και ένας αριθμός συστημάτων στήριξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για νούμερα τώρα αυτό σημαίνει ...870 εκατομμύρια λόγω της κρίσης και πάνω από 100 εκατομμύρια λόγω των συστημάτων στήριξης της ανανεώσιμης ενέργειας που έχουν ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση. Και τρίτο επιχείρημα είναι η, τρίτο πρόβλημα μάλλον είναι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των χωρών μελών βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου οι ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας και οι διασυνθέσεις είναι υψηλότερες από ποτέ, αλλά το επίπεδο συντονισμού είναι πολύ μακριά ακόμα από το επιθυμητό. Ένα και το καλύτερο παράδειγμα είναι η γερμανική ενεργή η στροφή δηλαδή στην ενέργεια, κάτι το οποίο έχει πολύ βαριές συνέπειες σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική, καθώς και σε γειτονικές χώρες. Και αυτό βεβαίως λόγω μιας απόφασης που λήφθηκε από την ε, κυβέρνηση αυτή χωρίς συντονισμό στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν έναν αριθμό προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και εξετάζοντας και πάλι όλη αυτή την ιστορία της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής αν τη δει κανείς από ψηλά αν μπορούμε να πούμε έτσι από το ελικόπτερο και αν συγκρίνεται την Ευρώπη με τις ΗΠΑ μπορείτε να πείτε ότι η δική μας παραγωγή ενέργειας αφενός γίνεται πιο βρώμικη, πιο δαπανηρή και οι παραγωγοί δεν εξασφαλίζουν σημαντικά κέρδη, ενώ στις ΗΠΑ γίνεται φτηνότερη παραγωγή ενέργειας, καθαρότερη και οι διάφορες δέκο εκεί βγάζουν και λεφτά. Εκεί λοιπόν πρόκειται για ένα πρόβλημα σχεδιασμού και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν η Business Europe έχει αναπτύξει 7 συστάσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ένα, και νομίζω ότι το είπα ήδη πριν, ίσως έχουμε ένα πρόβλημα, στην ισορροπία προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ανάμεσα στην πολιτική κλίματος και μείωση του κόστους. Εμείς προτείνουμε λοιπόν την εισαγωγή, την θέσπιση μάλλον στόχων για την αποτελεσματικότητα του κόστους και για την ασφάλεια προμηθειών. Βεβαίως και αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να αναλάβουμε τις ευθύνες όσον αφορά την ανάγκη προστασίας του κλίματος, νομίζω όμως ότι έχουμε δώσει υπερβολικό βάρος σε ένα πυλώνα, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να στηριχτούμε σε τρεις. Πρώτος, κόστος. Δεύτερο, ασφάλεια προμηθειών. Τρίτος, πυλώνας, βεβαίως, προστασία περιβάλλοντος και κλίματος. Αλλά πρέπει να βασιστούν και οι τρεις αυτοί πυλώνες σε ισότιμη βάση. Και εμείς νομίζουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει εφόσον βάλουμε ξεκάθαρους στόχους για μείωση του κόστους και ιδίως στην ανάγκη μείωσης του κενού που έχουμε στην αποδοτικότητα του κόστους σε σύγκριση με αυτό που έχουν οι ανταγωνιστές μας. Δεύτερο, και νομίζω ότι πολλοί εδώ τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα πρέπει να έχουμε τρεις στόχους, αλλά έναν στόχο μείωσης των ε, διοξιδίων του άνθρακος. Γιατί καμιά φορά οι άλλοι στόχοι προκαλούν στρεβλώσεις και είναι καλύτερα να δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα για να δοθεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα δηλαδή στους επενδυτές για να υπάρξει ασφάλεια για τις επενδύσει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν εκτιμούμε την υψηλή αξία των ε, ανανεώσιμων ενεργειών, σημαίνει όμως ότι δεν θέλουμε να βλέπουμε διαρκείς επιδοτήσεις υπέρ των ενεργειών αυτών. Να δοθεί ε, στήριξη στα αρχικά στέδια για να προσεγγίσουν την αγορά, όχι όμως πλέον σε ενέργειες οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ μακριά από την αγορά. Πάλι παράδειγμα από τη Γερμανία. Οι υπολογισμοί λένε ότι η μείωση ενός τόνου διοξιδίου του άνθρακος στη Γερμανία μέσω ηλιακών ε, πινάκων κοστίζει 600 ευρώ. Ακόμα δηλαδή και στους 30 να φτάσει ο τόνος του αερίου πάλι θα είναι 20 φορές παραπάνω η επιδότηση. Ποτέ δεν μπορεί λοιπόν να μπει αυτό σε ένα ορθολογικό σύστημα και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Όπως είπα, θα θεσπίζαμε έναν ενιαίο στόχο για την μείωση των εκπομπών που θα πρέπει να είναι κατάλληλος όσον αφορά και τους στόχους των άλλων τμήματων του πλανήτη. Δηλαδή, αν δείτε την εξέλιξη μέχρι τώρα, θα δείτε ότι ναι, μεν η Ευρώπη έχει κάνει πολλά ήδη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσει. Πρώτα πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε αναλάβει, μείωση, δηλαδή κατά 20% το 2020. Δεύτερο, είμαστε και έτοιμοι να στηρίξουμε και άλλο στόχο πέραν του 2020 για το 2030. Εάν δεν γίνει τίποτα, λέμε εμείς, στο υπόλοιπο του κόσμου. Αυτό δεν είναι αυτονόητο και συζητείται πολύ έντονα στην εκλογική μου περιφέρεια. Αλλά εμείς εμένουμε στο πρόγραμμα ETS της εμπορίας δηλαδή των ε, εκπομπών γιατί θεωρούμε ότι είναι το καλύτερο σύστημα. Αλλά βέβαια θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις φιλοδοξίες μας σε αυτά που μπορούν να τα αποκριθούν και οι άλλοι. Δεν θα μπορέσουμε να σώσουμε τον κόσμο μόνοι μας, τον πλανήτη μόνοι μας στις παγκόσμιες εκπομπές το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Υπήρου είναι 11%. Ενώ αυξάνεται σε όλα τα άλλα μέρη του κόσμου, σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Και για το 2030 το ποσοστό συμμετοχής μας θα είναι περίπου 4,5%. Αυτό αναμένεται τουλάχιστον. Ακόμα δηλαδή και αν εμείς μειώσουμε στο 0 τις εκπομπές μας, πάλι δεν πρόκειται να ανατραπεί η εξέλιξη αυτή σε ολόκληρο τον κόσμο. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε του στόχου μα. Αλλά πρέπει να ξανασκεφτούμε τη στρατηγική που έχουμε στήσει μέχρι τώρα. Και αυτή η ηγεσία δια του παραδείγματο, όπω είπαμε, η πρωτοπορία δια του παραδείγματο, δεν αποδίδει τα αποτελέσματα που θα θέλαμε να δούμε που θα ήταν μια φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία. Αυτό που είδαμε ωστόσο τελευταία και χαίρομαι γιατί για πρώτη φορά από την επιχειρηματική κοινότητα είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις με τους διαπραγματευτές. Αυτά που είδαμε στη Βαρσοβία όμως δεν κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. Είδαμε Ινδία και Κίνα πολύ διστακτικέ. είδαμε την Ιαπωνία ε, λίγο πολύ να, να περνάει από το μείον 25 στο συν 3 λένε μείον 5 αλλά σε διαφορετικά χρόνια. Άρα δηλαδή συνολικά μία απόκληση της τάξης του 28%. Εμείς θέλουμε να δούμε λοιπόν ένα φιλόδοξο στόχο. Να δούμε στόχο που να μπορεί να υποστηριχθεί αλλά που να είναι ρεαλιστικός. Και όπως λέμε μείον 40 δεν είναι ρεαλιστικό. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Και είπαμε ότι πρέπει να είναι και προσαρμοζόμενος ή προσαρμοστός ο στόχος, αναλόγως της πορείας των διαπραγματεύσεων. Εάν περισσότερες χώρες από ό,τι περιμένουμε τώρα ε, εμφανιστούν ικανές να μπουν σε μια παγκόσμια συμφωνία, τότε μπορούμε να ανεβάσουμε τον στόχο σε πιο ψηφιλόδοξα επίπεδα. Αν όχι όμως, τότε πρέπει να έχουμε την ικανότητα να μειώσουμε τους στόχους μας. Ή δε μη θα κάνουμε το ίδιο λάθος που κάναμε στην Κοπενχάγη και που δεν νομίζω ότι ισχυρίζεται κανείς ήταν μεγάλη επιτυχία. Είπα λοιπόν ήδη ότι θέλουμε να διατηρηθεί το σύστημα ETS της εμπορίας των ε, εκπομπών δηλαδή ως θεμέλιος λίθος γιατί ναι μεν έχει προβλήματα ωστόσο εμπεριέχει ακόμα πολύ αξία διότι είναι ένα σύστημα αγορακεντρικό και δεν αποκλείω στο μέλλον μετά το 2020 να υπάρχει και κάποιο περιθώριο για την θέσπιση ενός μηχανισμού που εάν έχουμε διαφορετικές εξελίξεις στην αγορά, δεν το λέω ότι θα γίνει αυτό, ε, το σύστημα να είναι προβλεπτό, διαφανές και όχι να βασίζεται σε βραχυπρόθεσμες πολιτικούς ελιγμούς. Όπως είπα, ε, είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όσον αφορά τις επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες ενέργειες. Θα θέλαμε αυτές σταδιακά να καταργηθούν Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι υπάρχει και ανάγκη ασφάλειας των επενδύσεων και ότι δεν μπορεί αυτές οι επιδοτήσεις να καταργηθούν από μια μέρα στην άλλη. Είδαμε όμως ότι έχουν στρεβλωτικό χαρακτήρα, ότι θέλουμε να δούμε η υποστήριξη στα αρχικά σχέδια μιας νέας τεχνολογίας, όχι όμως διαρκείς επιδοτήσεις. Επανέρχομαι τώρα στο συντονισμό. Νομίζουμε ότι θα χρειαστούμε ένα υποχρεωτικό σύστημα συντονισμού, έφερα το παράδειγμα πριν της γερμανικής τροφής στην ενέργεια, θα χρειαστεί τουλάχιστον υποχρεωτική διαβούλευση. Θα παραμείνει βέβαια αρμοδιότητα των χωρών μελών, αυτό δεν το αμφισβητούμε, αλλά αυτό που ζητούμε εδώ δεν είναι περισσότερη Ευρώπη, είναι καλύτερη Ευρώπη. Και χρειάζεται πραγματική ε, και υπάρχει μάλλον, μάλλον πραγματική ανάγκη καλύτερου συντονισμού. Άλλο θέμα κατά τη γνώμη μου σημαντικό, όταν λέω ότι το σύστημα ETS είναι το σωστό σύστημα, πρέπει να θυμηθούμε ότι σχεδιάστηκε για να είναι σύστημα βασισμένο στην αγορά και όχι να έχει δημοσιονομικό χαρακτήρα, δηλαδή ε, παρεμβάσεις δημοσιονομικές ενώ πολύ συχνά βασίζεται σε συμμαχίες, συνεργασίες με τα Υπουργεία Οικονομικών. Τουλάχιστον σε ορισμένες χώρες μέλη έχει φτάσει να είναι σχεδόν δημοσιονομικό εργαλείο. Ενώ ο λόγος που σχεδιάστηκε ήταν ακριβώς να μην παίζει το ρόλο δημοσιονομικού εργαλείου. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι τα χρήματα που εισπράττονται από το ETS θα πρέπει 100% να επανεπενδύονται στη βιομηχανία. Είτε μέσω αποζημιώσεων για να παραμείνει ανταγωνιστική στο παγκόσμιο επίπεδο, είτε πιο σημαντικό ακόμα, με άμεσες επενδύσεις σε αλλαγές στην οικονομία. Με άμεσες επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη για νέες τεχνολογίες που θα χρειαστούμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους ποθητούς σκοπούς. Και τέλος, επίσης πολύ σημαντικό, πολύ πολύ σημαντικό, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διαφοροποιήσουμε τις πηγές ενέργειάς μας. Αυτό βεβαίως συνεπάγεται και διαφοροποίηση των δυνατοτήτων, αλλά και καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων δυνατοτήτων. Μέσα σε αυτές που διαθέτουμε δηλαδή ήδη, διαφοροποίηση και μεταξύ αυτών και σχιστολιθικό αέριο. Τα είπα και πρόσφατα όταν, ε, είχα, όταν έλαβα το λόγο στην ε, συνάντηση Ανατολικής Γειτονίας, είδαμε τελευταία ότι αυτό οφείλουμε να το κάνουμε και για στρατηγικούς λόγους. Γνωρίζουμε ότι το αέριο θα παίξει μείζωνα ρόλο, τελειώνω σχεδόν, τελειώνω, θα παίξει μείζονα ρόλο το αέριο λοιπόν όπως είπα. Γνωρίζουμε ότι οι παραδοσιακές μας πηγές εξαντλούνται, γι' αυτό και πρέπει να διερευνήσουμε τις εναλλακτικέ πηγές και το σχιστολιτικό αέριο είναι μια εναλλακτική πηγή και δεν πρέπει να αυτοαποκλειστούμε από αυτή τη δυνατότητα. Τελειώνοντας λοιπόν θεωρώ ότι είναι σημαντικό να σχεδιάσουμε σωστά την πολιτική αυτή είναι σημαντικό να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος, του κλίματος κτλ. Αλλά δεν θα φτάσουν. Βεβαίω χρειαζόμαστε και πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σωστές ε, δεξιοτεχνίες και ικανότητες, άνοιγμα των αγορών και βεβαίω και πιο ευέλικτες αγορές εργασίας. Αυτό είναι όμως διαφορετική ιστορία. Ανάμεσα σε αυτά θα δούμε βεβαίω και ότι οι ενεργειακές πολιτικές είναι το κύριο Θεμέλιο. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας και για την προσοχή που χαρίσατε στα λόγια μου. Ευχαριστώ πολύ. Και Μπαγιά, πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Βεβαίως ότι θα ακολουθήσουν πολλές ερωτήσεις, διότι παρουσιάσετε μια εντελώς διαφορετική θέση. Και ο Σταγιάννη δεν έχει έρθει ακόμη. Οπότε, λόγος τον καθηγητή από τον Ιτρέχτη, ο κύριος Μπλοχ, θα μας μιλήσει για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και για εμπορικό ισοζύγιο. Ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας παρουσιάσω εντάχει τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και το μέλλον του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να θέξω τρία ζητήματα η συνεισφορά των ενεργειών αυτών ως το 2030. Δεύτερον, κάτι που είναι πολύ συζητημένο, πώς ενσωματώνουμε τις ανανεώσιμες το ηλεκτρικό μας δίκτυο και πώς θα ενθαρρύνουμε τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών. Σε ποιο βαθμό μπορούν να συνεισφέρουν οι ανανεώσιμες ε, πηγές το 2030 για να απαντήσουμε την ερώτηση αυτή. Κατασκευάσαμε ένα ευρέως παγκοσμίως θα λέγα χρησιμοποιούμενο μοντέλο το οποίο λαμβάνει υπόψη του τεχνικές, οικονομικές και άλλες παραμέτρους και περιορισμούς. Δεν θα επισέλθω στις λεπτομέρειες του μοντέλου. Θα σας παρουσιάσω τα κυριότερα αποτελέσματα. Εδώ βλέπετε, όπως προκύπτει σαφώς, το σενάριο ως το 2030. Μπορεί να τα διαβάζετε όλοι σας ε, ειδικά στο βάθος της αίθουσας. Να σας πω δύο λόγια όμως. Πάνω πάνω είναι η συνολική χρήση ενέργειας. Βλέπετε ότι πέφτει χάρη στην πιο ποδοτική χρήση της ε, ενέργειας. Αυτό είναι και το βασικό μας σενάριο αν θέλετε. Δεν θα με το θέμα αυτό, θα σας το παρουσιάσει ο επόμενο ομιλητή. Βλέπετε εδώ και τη συνεισφορά των ανανεωσιμών. Συμπέρασμα, μπορούμε να πετύχουμε ένα 40% το 2030. Δεν ε, προφανές, αλλά δεν είναι και πολύ δύσκολο. Εξαρτάται τι στόχους έχουμε και που θέλουμε να πάμε. Αν δούμε τώρα την κατανομή των διαφορών πηγών βλέπετε μεγάλη ποικιλία, μεγάλη διασπόρα διαφορών πηγών που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν προς την επίτευξη του στόχου. Κάτω με γαλάζιο βλέπετε την αιωλική ενέργεια, επίγεια και παράκτεια, Μετά με κίτρινο και πορτοκαλί διάφορες μορφές ηλιακής ενέργειας, κυρίως για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και εν μέρη, για παραγωγή θερμότητας. Τα υδροελεκτρικά είναι σχετικά σταθερά και ως προς την γεωθερμία ένα μικρό ποσοστό και κάποιες συνεισφορές από βιομάζα. Εδώ μιλάμε κυρίως για τα απόβλητα αλλά και πολύματα ξύλου. Όμως συμπεριλαμβάνουμε και πολύματα καλλιεργιών. Ένα ποικίλο μείγμα λοιπόν. Η παραγωγή ηλεκτρισμού καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος τις ε, απορρόφησης ενέργειας. Το θέμα είναι λοιπόν να μετατρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερη ηλιακή και ολική σε ηλεκτρισμό. Πάρω στο 40% παραλαμβάνω είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Φυσικά αυτά ποικίλουν από το μέσα τομέα. Βλέπετε τα κτίρια αριστερά επάνω, λίγο λιγότερο στην βιομηχανία. Εδώ μιλάμε και για ηλεκτρισμό και για ενέργεια και στις μεταφορές δεξιά επάνω. Εδώ βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση, αριθμό που θα καμφθεί μετά. Συνεπώς, αναμένουμε συνεισφορά από όλους τους τομείς. Ας δούμε τώρα και τα κόστη. Η ανωγραμμή γραμμή είναι επενδύσεις. Τι πρέπει να επενδύουμε κάθε χρόνο για να επιτευχθεί ο στόχος. Βλέπετε ότι έχουμε υψηλές επενδύσεις. Πρέπει να επενδύουμε τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ μας κάθε χρόνο για να μπορέσουμε να κινηθούμε προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Όχι μόνο για τις ανανεώσιμες αλλά και για τα μέτρα αποδρικής χρήσης της ενέργειας, για την ενίσχυση των δικτύων, για έρευνα και ανάπτυξη. Ένα σύνολο λοιπόν μέτρων που απαιτούν αυτές τις επενδύσεις. Δεν ακριβώς λοιπόν. Κόστος είναι επενδύσεις. Εξοικονομήσεις κάτω η μπλε γραμμή στικτή γραμμή. Εδώ έχουμε μείωση. Είναι το αρνητικό κόστος χάρη στην αποφυγή χρήσης δηλαδή ορυκτών καυσίμων και στην πράσινη γραμμή. Βλέπετε ότι κατά την πρώτη μία μισή περίπου δεκαετία έχουμε καθαρές επενδύσεις. Εν συνεχεία έχουμε τα καθαρά ωφέλη. Το κόστος αυτό βεβαίω, ο πολιτισμός τουλάχιστον βασίζεται σε κάποιες παραμέτρους όπως η τιμή του πετρελαίου αλλά, ή των δικαιωμάτων εκπομπών. Αυτό μια άλλη ιστορία. Θα μπορούσαν σε αρτήσει διαφορετικών τιμών τα ωφέλη να είναι ακόμα μεγαλύτερα. Πετυχαίνουμε μεγάλες επίσης μειώσεις των ε, εκπομπών το 2030. Οι εκπομπές όχι των αερίων θερμοκηπίου αλλά του διοξιδίου ε, του άνθρακα θα είναι μισές, θα είναι κατά 50% χαμηλότερες από τις εκπομπές το 1990. Επόμενο ερώτημα, πώς θα σωματωθούν οι ανανεώσιμες το ηλεκτρικό μας δίκτυο. Και πάλι όχι πολλές λεπτομέρειες, μερικά σενάρια αν θέλετε. Καταρχήν μια εικόνα που αποτυπώνει το σημερινό ηλεκτρικό δίκτυο, τη σημερινή ηλεκτροπαραγωγή. Αυτό είναι το κλασικό παραδοσιακό σενάριο για την Γερμανία. Μια ημέρα του χειμώνα, στην μια εβδομάδα του χειμώνα μάλλον στη Γερμανία. Παραδοσιακή κατανομή. Εδώ βλέπετε ότι η παραγωγή, την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στη Γερμανία επί μια εβδομάδα. Οι καθημερινές διακυμάνσει ε, λιγότερη κατανάλωση τη νύχτα βεβαίως και πάνω βλέπετε ότι ένα μέρος αυτής της ενέργειας παράγεται από τον άνεμο. Κυλιακή βεβαίως. Και βλέπετε την ανάλυση των πηγών που χρησιμοποιούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έχετε δει νομίζω αυτά. Ξεκινάει κανείς με την φθηνότερη ενέργεια, μετά τις ανανεώσιμες, με το μικρότερο οριακό κόστος, πυρηνική ενέργεια, το κόκκινο βεβαίως, μετά ο λιγνίτης, ο καφέ άνθρακας, ο λιθάνθρακας μετά με μαύρο, το πορτοκαλί είναι το φυσικό αέριο. Είναι το κλασικό αν θέλετε σενάριο. Έτσι λειτουργούν τα εργοστασιά μας, τα οποία κλείνουν τη νύχτα, μειώνουν τη δραστηριότητά τους και παρέχονται το πρωί. Αυτά ίσχυαν και πριν από 10 χρόνια. Όμως, μια τυπική χειμωνιάτικη μέρα που δεν έχουμε αρκετή ολική ηλιακή ενέργεια στη Γερμανία. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε τώρα στο καλοκαίρι. Μια εβδομάδα του Ιουνίου, μια συγκεκριμένη εβδομάδα του 2013. Τι βλέπουμε εδώ. Τελείως διαφορετική εικόνα. Βλέπετε εδώ πολύ ηλιακή ενέργεια, η οποία παράγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό το γνωρίζουν όλες οι εταιρείε. Δεν υπάρχει πολλή χώρος, να το πω έτσι, για το φυσικό αέριο. Δεν είναι δηλαδή απαραίτητο. Τα ηλεκτρικά εργοστάσια που και είναι λιθάνθρακα μπορούν να κλείσουν σχεδόν και μπορούμε να μειώσουμε και την παραγωγή από πυρηνικά εργοστάσια. Αξιοσημείωτο εδώ είναι πρώτον το εξή, ότι το επόμενον το πλεονασματικό φορτίο είναι πολύ πιο σταθερό από ό,τι ήταν παλιά. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ του φορτίου της μέρας και του φορτίου της νύχτας είναι πολύ μικρότερη και δεύτερον η ανάπτυξη με πράσινο των της παραγωγής λειτουργού ρεύματος που ανανέωσουμε είναι σχετικά ομα, ομαλότερη, πιο σταθερή. Και αυτό γιατί παλιά είχαμε διαφορές, μεταβολές μάλλον, απρόβλητες ε, μεταβολές στην παραγωγή αιωλικής ενέργειας με το δεκάλεπτο. Αυτό όμως αλλάζει πλέον συνολικά για τις ανανεώσιμες. Τιμές. Παλιά οι τιμές τι ενέργειε από ανανεώσιμε ήταν πολύ ψηλέ. Είχαμε και διαφορά μεταξύ νύχτα και ημέρα. Χάρη στην αιωλική και την ηλιακή Όμω βλέπετε ότι οι τιμέ έπεσαν. Έτσι έχει μειωθεί και το οριακό κόστος στη Γερμανία συγκεκριμένα σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτό είναι μια τάση που εξαπλώνεται και στην Ολλανδία και σε άλλες γειτονικέ χώρες οι οποίε μάλιστα γειτονικέ χώρε ε, διαμαρτύρονται για τι χαμηλέ τιμέ στην ενέργεια στη Γερμανία. Ε, σε μερικέ περιπτώσει μάλιστα είχαμε και αρνητικέ τιμέ όπω βλέπετε δεξιά στο διάγραμμα. Τι γίνεται λοιπόν όσο μπαίνει περισσότερο ηλιακή ενέργεια στην εικόνα. Παλιά όπως είπα ήταν κάπως έτσι η κατάσταση, είχαμε τις γνωστές εχμές. Τώρα όμως έχουμε το πρότυπο του μοντέλου της καμήλες Δύο ύβους, δύο κορυφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ως εκ του συνδυασμού της παραγωγής και της, ε, του μοντέλου της κατανάλωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό πειράζει λοιπόν τα εργοστάσια, τα οποία λειτουργούν με πολύ διαφορετικό τρόπο σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Η Γερμανία και άλλες χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο έως και να διπλασιάσουν το ποσοστό των ανανεωσίμων στην παραγωγή τους. Βεβαίως η πρόκληση είναι η εξορρόπηση προσφοράς και ζήτησης. Και το λόγω της απαιτούμενης ευελιξίας. Οι εναλλακτικές λύσεις, αν θέλετε, είναι αυτές που βλέπετε εδώ. Πώς λειτουργεί το σύστημα. Καταρχήν χρειαζόμαστε ευελιξίες προς την παραγωγή, την προσφορά. Εκεί συμμετέχουν όλα τα εργοστάσια, όχι μόνο τα συμβατικά, αλλά και αυτά που παράγουν ανανόσιμη ενέργεια. Και εκεί χρειάζεται ευελιξία. Ευτυχώς στην εξόρροπηση του δικτύου συμμετέχουν τώρα πια και η ολική και η ηλιακή ενέργεια. Η ζήτηση και αυτή μεταβάλλεται. Εδώ έχουμε πολλές δυνατότητες. Μάλιστα έχουμε εξελίξεις οι οποίες θα διαμορφώσουν διαφορετικά το μέλλον, ηλεκτρικά αυτοκίνητα για παράδειγμα. Γι' αυτό θα επηρεάσει τη ζήτηση της ενέργειας. Εάν οι τιμές πέσουν εκεί, το φαινόμενο θα ενταθεί. Προς το παρόν, η πιο σημαντική παράμετρο σαν είναι το δίκτυο. Εκεί Έχουμε μεγάλα αποθέματα ευελιξίας. Χρησιμοποιούμε δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα εδώ, ένα ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο παράγεται αλλού. Η επέκταση του δικτύου εδώ θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο. Και τέλος η αποθήκευση ενέργειας. Δεν το πολύ συζητούμε, αλλά από οικονομικής απόψεως είναι μια δυνατότητα, όχι πολύ σημαντική όμω. τουλάχιστον βράχει πρόθεσμα, ειδικά όσον αφορά το φυσικό αέριο για παράδειγμα, ίσω σε 20 χρόνια από τώρα. Προς το παρόν όμως δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά από αυτήν την άποψη. Η ανάλυση αυτή αφορά την Γερμανία και είναι αρκετά λεπτομερή. Βασίζεται στο, στην υπόθεση εργασία ότι το δίκτυο δεν θα επεκταθεί το δίκτυο διανομής ως το 30. Ακόμη και έτσι όμως η Γερμανία δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα ως το 2030 με τα παρόντα τη σημερινή εργοστάσια και το σημερινό δίκτυο. Φυσικά θα ήταν πιο φθηνό το κόστος, εάν το δίκτυο έχει επεκταθεί, θα μας επέτρεπε κάποιους εξορθολογισμούς. Άρα η επέκταση των δικτύων εν είναι ένα κρίσιμο θέμα. Αυτά λίγο πολύ μπορούμε να κάνουμε. Αυτά ως μια γενική επισκόπηση. Υπάρχουν πολλές, πολλοί τρόποι να γίνει πιο ευέλικτο το σύστημα, το δίκτυο, υπάρχουν προκλήσεις, όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν. Τέλος, τρίτο ζήτημα, το τρίτο που ήθελα να θίξω. Έχω λίγο χρόνο, οπότε θα το περάσω λίγο γρήγορα. Πώς προάγουμε τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Εδώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Όλες αξιοποιούνται στην Ευρώπη. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι έχουμε Προσωστώσεις, έχουμε ειδικέ τιμές προμήθειας στο δίκτυο και άλλου είδους κίνητρα έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε την παραγωγή ανανεωσίμων μορφών ενέργειας. Θα έλεγα ότι η σύγκληση εδώ είναι ένα σημαντικό θέμα και βλέπετε κάποια σύγκληση στις μέρες μας. Όλο και λιγότερες χώρες χρησιμοποιούν ποσοστώσεις, κάποιες ε, άλλες θεσπίζουν ειδικές τιμές συνεισφοράς ε, στο δίκτυο ή αγοράς από το δίκτυο. Εδώ αναλύουμε τα επιμέρους, τα διαφορετικά συστήματα ανά την Ευρώπη και ε, ποια συστήματα αποδίδουν και ποια όχι. Καταγράφουμε ορισμένα βασικά χρήσιμα συμπεράσματα. Ε, και τα οποία ανατρέπουν κάποιους παραδοσιακούς, ε, κάποια παραδοσιακά πιστεύω. Ότι η εναρμόνιση για παράδειγμα λύνει τα πάντα. Χρειάζεται αλλά προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Λοιπόν, τα βασικά μας συμπεράσματα από την ανάλυση είναι πρώτον, αν και αυτό ακούγεται σε πολλές χώρες, το γνωρίζουμε, χρειάζεται ένα αξιόπιστο πλαίσιο, σύστημα υποστήριξης με διάρκεια, ένα σταθερό σύστημα. Γιατί αλλιώς ανατρέπεται η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Δεύτερον, πρέπει να λάβουμε υπόψη τους ε, κινδύνου για τι επενδύσεις. Τα συστήματα μπορούν να σχεδιαστούν με διαφορετικούς τρόπους. Κάποια συστήματα όμως ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους για του επενδυτέ. Και ως εκ τούτου, και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σε, οδηγούν σε υψηλότερο κόστος της ενέργειας. Το θέμα εδώ είναι να μειώσουμε και το κόστος της ενέργειας. Και τέλος, πετυχαίνει κανείς το μικρότερο κόστος όταν προσαρμόζει την, τις επιδοτήσεις στην τεχνολογία και στην αγορά. Ήδη έχει μειωθεί το κόστος της υποστήριξης, της ενίσχυσης των ανανεωσίμων τα τελευταία χρόνια και τούτο λόγω μάλλον χάρη στην προσαρμογή τη εξελίξεις. Ένα ε, κατακλείδη, είναι δυνατόν να αυξήσουμε τη συμμετοχή των ανανεωσίμων. Υπάρχουν προκλήσεις, μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με τρόπο ρεαλιστικό και εν τέλει όσον αφορά τις ενισχύσεις, την επιδότηση αν θέλετε των ανανεωσίμων, χρειαζόμαστε μια προσαρμοσμένη ευέλικτη προσέγγιση, η οποία από οικονομική άποψη είναι πιο σε σύγκριση με μια συνολική προσέγγιση προ τον ίδιο ακριβώ στόχο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Έφτασε και ο κύριος Ταγιάννη, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαίρομαι πολύ που παρευρίσκεστε εδώ και σας ευχαριστώ που αφιέρωσατε χρόνο για αυτή την συνεδρίαση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο, ο οποίος θα αναφερθεί στο θέμα των ενεργειακών πηγών για μια αντιγωνιστική βιομηχανία. Ευχαριστώ, θα μιλήσω τη μητρική μου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ από τα Εθνικά Κοινοβούλια, η σημερινή συνεδρίαση είναι πάρα πολύ σημαντική για να εντάξουμε το θέμα της ενέργειας στο πλαίσιο της επιστροφής σε μια σύγχρονη και ανταγωνιστική βιομηχανική πολιτική. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ένα στόχο 20% του καθαρίστου χώρου προϊόντος ε, πριν τα τέλη του 2020, που να προέρχεται από τη μεταπαιδική βιομηχανία. Εμείς ε, θα παρουσιάσουμε σε λίγες εβδομάδες μία ανακοίνωση η οποία θα αποτελέσει και σημαντική συνεισφορά για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου όπου θα συζητηθεί το θέμα της ανταγωνιστικότητας ε, του βιομηχανικού συστήματος. Ε, και εγώ νομίζω ότι μαζί με το Fiscal Compact ε, χρειάζεται δηλαδή πέρα από το σύμφωνο για τη φορολογία και ένα σύμφωνο για τη βιομηχανία προκειμένου να δώσουμε μία όθηση στην πραγματική οικονομία. Όμως για να έχουμε μία νέα και σύγχρονη βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ορισμένα σημαντικά θέματα να επικεντρώσουμε τις προσπαθίες μας σε ορισμένες δράσεις, νέες τεχνολογίες, καινοτομία, πρόσβαση στην αγορά, διεθνοποίηση, πρόσβαση στα κεφάλαια, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στις δεξιότητες, στην κατάρτιση. Αλλά υπάρχει και ένας θεμελιώδης πυλώνας της ενεργειακής πολιτικής. Δεν είναι τυχαίο που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου ανέθεσε στην Κομισιόν το καθήκον να προετοιμάσει και ενόψεις του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου ένα έγγραφο το οποίο θα μπορούσε να καταδείξει ποιος είναι ο αντίκτυπος της ενεργειακής πολιτικής επί της βιομηχανικής πολιτικής. Συνεργαζόμαστε με τον Επίτροπο Έτιγκερ και το έργο μας θα παρουσιαστεί πριν από την υλοποίηση του Συμβουλίου. Έχουμε φιλόδοξους στόχους ήδη ε, με ε, τους ε, με τις διαδικασίες με για το 2050, κάτι που θα δώσει μεγάλη όθηση στην οικονομία μας και το ενδιάμεσο πλαίσιο για την ενέργεια και το κλίμα το 2030 αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά χρειαζόμαστε κατάλληλες πολιτικές απαντήσεις μέσω πρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα για να διασφαλίσουμε ότι φιλόδοξοι στόχοι θα επιτευχθούν με το λιγότερο κόστος για την κοινωνία και τη βιομηχανία. Επίσης πρέπει να έχουμε μια συνεχή προσέγγιση μεταξύ των πολιτικών δράσεων έχοντας κατά νου ότι η προτεραιότητά μας είναι να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως έναντι του υπόλοιπου κόσμου έχοντας υψηλή ενεργεία και μια βιομηχανική βάση η οποία συνεχώς συρρυκνώνεται πρέπει να εκμεταλλευτούμε ως δυνατόν καλύτερα όλες τις οικονομικές και παραγωγικές ικανότητες που μας οδηγούν προς μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διεξοδίου του άνθρακα και αποτελεσματική ως προς τη χρήση των πόρων. Και επομένως είναι προτεραιότητα το θέμα του τιμών της ενέργειας. Είναι πάρα πολύ υψηλές στην Ευρώπη και έτσι χάνουμε ανταγωνιστικότητα. πληρώνουμε την ηλεκτρική ενέργεια πολύ πιο ακριβά από την Κίνα. Και το να παράγει κανείς με ένα τέτοιο κόστος σημαίνει πραγματικά ότι ε, ταξιδεύει με μόλιδο στα φτερά του, δηλαδή με πολύ μεγάλο βάρος. Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο σε όλους, ε, όμως ε, δεν είναι και εύκολο να βρεθούν οι λύσεις. Αναλύουμε το πιο πρόσφατα δεδομένα της, του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και προκύπτει ότι οι καταναλωτές στην Ευρώπη μαζί με τους Ιάπωνες πληρώνουν πάνω από το διπλό για ε, την ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση με το πόσο πληρώνουν οι καταναλωτές της Ηνωμένης Πολιτείας. Επίσης, έχουμε την τιμή του αερίου που είναι τρεις φορές χαμηλότερη εκεί και έχουμε και το σχεστολιθικό αέριο που πρέπει να αυστήσουμε την προσοχή μας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν αρκετά σαφές ζητά να προχωρήσουμε, να σημασούμε πρόοδο σε αυτό το θέμα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια ουδέτερη στάση απέναντι στο θέμα αυτό. Υπάρχουν ανησυχίες για το περιβάλλον, αλλά υπάρχουν και ανησυχίες οικονομικού και βιομηχανικού χαρακτήρα οι Ηνωμένε Πολιτείε προχωρούν στην παγκόσμια σκηνή χάρη στην ανταγωνιστικότητά τους που είναι καρπός του χαμηλού κόστους ε, της ενέργειας ε, επειδή χρησιμοποιούν σχιστολιθικό αέριο. Η Ευρώπη δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη το πρόβλημα αυτό. Να επαληθεύσει με επιστημονικό τρόπο, χωρίς προκαταλήψεις, υπέρ κατά, αν ε, θα προκληθούν ε, ζημίες στο περιβάλλον από την εξόρυξη του σχιστολιθικού αερίου για να δούμε αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως πηγή ενέργειας για τις επιχειρήσεις μας. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα μέσα που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας ε, για να ασκήσουμε την ενεργειακή πολιτική. Και υπάρχει ένα αίτημα από τα κράτη-μέλη να μην ε, είμαστε διστακτικοί στο αυτό και ο κύριος Κάμερον ε, έστειλε μια επιστολή και στον πρόεδρο της Κομισιόν ζητώντας να αναλυφθεί μια ισχυρή δράση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ ζητώ να γίνει μια ευφυής και προσεκτική ανάλυση για τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και στη συνέχεια να λάβουμε μια απόφαση. γιατί μπορεί το τίμημα να είναι πολύ ψηλό. Κατόπιν υπάρχουν μη ενεργητικές συνιστώσεις, όπως είναι οι φόροι, το κόστος της διανομής και η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συνεχώς αυξάνονται και μπορεί σήμερα να ε, φτάσουν στο 40 έως το 45% της τελικής τιμής ε, που πληρώνουν οι βιομηχανικοί, οι εταιρείε, η βιομηχανία. Έτσι λοιπόν υπάρχει πολύ ισχυρός αντίκτυπος όλων αυτών στην τιμή της ενέργειας. Όπως σας είπα, η ενέργεια είναι σημαντική, το, το κόστος είναι σημαντικό όχι μόνο για την ενεργοβόριο βιομηχανία, αλλά και για άλλες βιομηχανίες, αλλά και για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει το να υποστηρίξουμε την, ενεργοβόρο βιομηχανία στην περίπτωση αυτή είναι κάτι απαραίτητο και συνεισφορούμε ότι η συνεισφορά τους ε, σε ό,τι φορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι κάτι πολύ σχετικό, αλλά αν δούμε και τη στρατηγική τους θέση, το στρατηγικό ρόλο που έχουν εντός της αλυσίδας αξίας, ενισχύεται αυτό. Έχουμε δηλαδή πολύ ψηλό κόστος απέναντί μας, αλλά βλέπουμε και κάποια πραγματικότητα βιομηχανική που είναι πολύ σημαντική για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του ψηλού κόστους της ενέργειας, πολύ ψηλού ορισμένες φορές. Και φυσικά δεν θέλουμε να δούμε υπαναχώρηση σε αυτά τα είδη βιομηχανίας. Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι μια απάντηση, δηλαδή να μειώσουμε και το συναφές κόστος. Όμως όταν ε, οι αποφάσεις επενδύσεων περιλαμβάνουν και δαπανηρές λύσεις για σχέδια μεγάλης κλίμακας, αντιμετωπίζουμε νέα προβλήματα και έχουμε και την εναλλακτική λύση της μεταφοράς των εργοστασίων. Γιατί το κόστος, το μεγάλο κόστος της ενέργειας μπορεί να οθήσει τις ενεργοβόρες βιομηχανίες να πάνε να παράξουν πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν πρέπει να αναλύσουμε το κόστος και να το αξιολογήσουμε με ένα πολύ προσεκτικό τρόπο. Και θα πρέπει να προβούμε σε ένα καλύτερο συντονισμό των εθνικών πολιτικών και είναι και σημαντικό τα μέτρα παρακολούθησης ε, για τους τομείς που είναι ενεργοβόροι να αποφύγουν τη στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς και να δημιουργηθούν και κανόνες ίση για όλους σε παγκοσμίο επίπεδο. Τώρα μια μικρή παρέκκληση σε σχέση με τους κανόνες ε, για τον ανταγωνισμό που έχουν θεσπιστεί για να ευνοήσουν την εσωτερική αγορά και κατά την άποψή μου θα να ίσως να μην είναι κατάλληλη μπροστά σε μια κατάσταση που θα έχει μεταβληθεί. Γιατί η ενεργοβόρος βιομηχανία μας στη δεκαετία του 50 ουσιαστικά ανταγωνιζόταν, πρέπει σε ανταγωνισμό μόνο σε επίπεδο εσωτερική αγορά. Ενώ σήμερα, επειδή έχει αλλάξει εντελώ η γεωπολιτική κατάσταση, βλέπουμε ότι πρέπει να ανταγωνιστούμε με κάποιες πραγματικότητες ε, όπως ε, της Βραζιλίας, της Κίνας, της Ινδίας. Και επομένως ε, και οι κανόνες του ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι αντικείμενο αξιολόγησης. Σίγουρα δεν εγκαταλείπουμε την αξία του ανταγωνισμού, όμως η εφαρμογή της αρχής μέσω των κανόνων θα πρέπει ουσιαστικά να ακολουθεί και τους καιρούς μας. Κάτι άλλο σε σχέση με το κλίμα και την ποιότητα της ατμόσφαιρας για το 2020. Θέλουμε να επικεντρωθούμε σε όλες αυτές τις συνιστώσεις και να θέσουμε τέτοια επίπεδα φιλοδοξίας έτσι ώστε να αποφύγουμε την αύξηση των τιμών ενέργειας και τη διαφοροποίηση μεταξύ των τιμών της ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυρίων ανταγωνιστών της. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους από την ανασιώσιμες πηγές ενέργειας και τις μη συμβατικές και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη. η δική μας στρατηγική για την εκβιομηχάνηση τονίζει ακριβώς αυτές τις τύχες. Όταν μιλάμε για την εκβιομηχάνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνουμε λόγο και για μια πολιτική που θα έχει στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση και την έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακόμη και αν δεν θα είναι εύκολο, αλλά πρέπει να δρούμε πάντοτε έτσι ώστε πάντοτε στις εργασίες μας να λαμβάνετε υπόψη το θέμα της ενεργειακής εξοικονόμησης και ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο τμήμα της παραγωγής μας ε, καταστάθηκε στην Κίνα όπου η κύρια πηγή ενέργειας είναι ο άνθρακας και έτσι η Κίνα σήμερα είναι ε, υπεύθυνη για τις περισσότερες εκπομπές του άνθρακα σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη έχασε 300 δισεκατομμύρια ευρώ ε, στο επίπεδο της βιομηχανικής παραγωγής και από το 40% έπεσε στο 20% και πάντοτε ωφελήθηκε η Κίνα. Πέρα από τον Ατλαντικό τώρα, είπαμε ότι έχουμε το θέμα του σχιστολιτικού αερίου, το οποίο πραγματικά τροποποιεί το ενεργειακό μείγμα του Αμερικανικού συστήματος με μια συνεχή μείωση του κόστους της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι λοιπόν εμείς θα πρέπει να πράξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε το μελλοντικό ενεργειακό μείγμα να περιλαμβάνει στο σύνολό τους όλες τις ενεργειακές μας πηγές. Φυσικά το υψηλό κόστος της ενέργειας, όπως είπαμε και στην αρχή, γίνεται ένα κεντρικό τμήμα της πολιτικής της Ενωσής μας. Θα πρέπει να βρούμε μια ορθή ισορροπία για το θέμα του σχιστολιθικού αερίου. Θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις. Γιατί διαφορετικά το σχιστολιθικό αέριο είναι ένας από τους τομείς ε, προς διερεύνηση, αλλά αν δεν ε, προβούμε σε μια άμεση επέμβαση επί όλων αυτών των ενεργειακών μέσων, τότε υπάρχει κίνδυνος πτώσης της ανταγωνιστικότητας και η διαφορά του κόστου της ενέργειας θα καταστήσει το ευρωπαϊκό βιομηχανικό σύστημα πραγματικά αδύναμο. Όπως ε, είπα, πριν από τη Σύνοδο Κορφής του Φεβρουαρίου θα παρουσιάσουμε αυτή την έκθεση της Γενικής μου Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης του Επιτρόπου Έτιγκερ για να προβούμε σε μια συγκεκριμένη συνεισφορά. Σε ό,τι με αφορά, θεωρώ ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την επικοινομορφία του ενεργειακού μείγματος, τον αντίκτυπο των ε, επιδοτήσεων για τις ενώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό πρέπει να μελετηθεί λεπτομερώς και ιδίως εκεί όπου η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν άμεση ευθύνη για τη χρηματοδότηση του backup. Η Κομισιόν παρουσίασε τον περασμένο μήνα της κατευθυντήρης γραμμής για την εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων για τον τομέα ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι από αυτά εξαρτώνται οι επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα πριν λίγες μέρες στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Κατόπιν έχουμε και το θέμα της σταδιακής εξάλληψης της πυρηνικής ενέργειας και το να αποκλείσουμε τη χρήση μη συμβατικών πηγών ενέργειας στην Ένωση και αυτό θα δώσει ε, μια πλεονεκτική, θα βάλει σε πλεονεκτική κατάσταση στους ανταγωνιστές μας, μια αύξηση ε, τη συνεισφορά του Πέλεν στη μείωση των ε, αποθεμάτων ε, του άνθρακα είναι κάτι σημαντικό. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε να θέτουμε στο επίκεντρο της ανέσιμες πηγές, να βρούμε νέες λύσεις για τη μείωση του κόστους, να προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα των διασυνδέσεων σε διεθνές επίπεδο για να μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους του 2020. Επίσης, η ανάπτυξη των ενώσιμων πηγών ενέργειας ε, να μην συνεισφέρει μόνο, δεν συνεισφέρει μόνο στους στόχους ε, της Ευρώπης 2020, γιατί τα νέα μοντέλα τους πράσινου επιχειρήν αποτελούν νέες ευκαιρίες για τους επιχειρηματίες μας. Σήμερα παρουσίασα τα αποτελέσματα του Ευρωβαρομέτρου για το πώς οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οδεύουν προς ε, μια πιο πράσινη προσέγγιση. Όλες οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις έχουν επιλέξει μία οδό και για λόγους εξοικονόμησης αλλά και από πεποίθηση που τους οδηγεί σε ένα σύστημα που ρηπαίνει λιγότερο, ένα πιο πράσινο σύστημα. Αυτό αποτελεί κάτι πολύ σημαντικό για μας τους Ευρωπαίους, μια σημαντική τεχνογνωσία. Εγώ έχω παρακολουθήσει τις εξελίξεις ε, σε κάποιους τομείς, ιδίως ε, στον τομέα των υδάτων και στο Ιστρέλ και στην Κίνα, με μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των συνομιλητών των δύο αυτοχωρών, οι οποίοι έχουν εκτιμήσει την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία. Επομένως, όλο αυτό το έργο, όλη αυτή η δουλειά μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική για την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά θα πρέπει να είμαστε και πιο θεραλέοι στις επιλογές μας και να απαντήσουμε στις απαιτήσει της ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και πρέπει να δώσουμε την απάντηση περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια πραγματική αγορά ενέργειας. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτό πρέπει να γίνει αν θέλουμε το ενεργειακό μας σύστημα να είναι ένα μέσο που θα υποστηρίζει ισχυρά την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, με το στόχο πάντοτε να έχουμε ένα σύστημα που δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας για να ακούμε και από την κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ενέργειας και του επιχειρήν. Ο τελευταίος τώρα, ο μιλητής θα μιλήσει για την αποδοτικότητα της ενέργειας που είναι το σχιστολιτικό αέριο της Ευρώπης. Ο κύριος Μπόι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλες και όλους. Θέλω να σας πω πρώτα λίγα λόγια. Όχι τόσο για το, ίδιο σχιστολιστικό αερίο, αλλά για μια εναλλακτική επιλογή. Άκουσα τα σχόλια του κ. Ταγιάννη και συμφωνώ ότι η αποδοτικότητα είναι μια πιθανή εναλλακτική επιλογή. Για, για μένα και για πολλούς άλλους που δουλεύουμε στον τομέα αυτό είναι σωστό. Το πρωί συζητήσαμε τα προβλήματα αυξανόμενες τιμές, μείωση της ανταγωνιστικότητας, ο επικρεμάμενος κίνδυνος της αλλαγής του κλίματος και μέσα σε αυτά και η ανεργία. Πολλά προβλήματα προκαλούνται από τοπική ρήπανση οι περισσότερες πόλεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη παραβιάζουν τα όρια των εκπομπών, εκπέμπουν πολύ περισσότερες εκπομπές ρήπων από ό,τι θα επέτρεπαν οι συμφωνίες του ΠΟΕ. Υπάρχει λοιπόν και ένα πρόβλημα υγείας εκτός από όλα τα άλλα. Πώς να τα λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Εδώ νομίζω μετά από την συζήτηση του σημερινού πρωινού μπορούμε να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα ότι ε, δεν είναι τόσο το θέμα των τιμών της ενέργειας όσο του κόστους της ενέργειας και του αριθμού των πόρων που χρησιμοποιεί κανείς. Τι σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Δεν σημαίνει μονάχα φθηνά προϊόντα σημαίνει ποιότητα, σημαίνει κατάλληλα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, πολλά πράγματα που συναπαρτίζουν την ανταγωνιστικότητα. Και νομίζω ότι συγκρίνουμε τώρα λίγο πολύ στις ιδέες αυτές και βέβαια πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος, να πετύχουμε ανάπτυξη που αυτή είναι που θα οδηγήσει σε επενδύσεις γιατί το ένα θρέφει το άλλο να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και του κεφαλαίου και της εργασίας να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της υγείας και για να γίνει αυτό πρέπει να μειώσουμε τη ρήπανση. Αυτό που προσπαθώ να πω με τα λόγια αυτά είναι ότι δουλεύοντας πάνω στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και χρησιμοποιώντας την ενιαία αγορά για να ολοκληρώσουμε και την αγορά αποδοτικότητας της ενέργειας που είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της αγοράς, μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ στην κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων που ανέφερα. Ακούσαμε από τον καθηγητή κύριο Μπλοκ για τις βιώσιμες ανα, ε, ανανεώσιμες ενέργειες που υπάρχουν, ηλιακή, αιωλική, γεωθερμική, παλιροϊκή ενέργεια, γιατί έχουμε τέτοια τα παλιροϊκά κύματα διαρκώς. Αυτά είναι το μέλλον. Το σχιστολιθικό αέριο, όπως είπε ο Επίτροπος Ταγιάννη, πρέπει να το εξετάσουμε προσεκτικά. Όμως έχουμε δείξει ήδη ότι δεν πρόκειται για βιώσιμη εναλλακτική επιλογή. Οι ΕΠΑ Πολιτείε έχουν ειδικέ συνθήκε εκεί. Αν πετάξετε πάνω από τι ΕΠΑ Πολιτείε, θα δείτε ότι οι μισέ δυτικέ πολιτείε είναι στην ουσία ακατοίκητες. το να πάνε εκεί να βγάλουν με τις ε, διάφορες ε, διαδικασίες που ρηπαίνουν. Το συστολιστικό αέριο είναι κάτι απλό. Στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης δεν θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο. Τέλος, όταν μιλεί κανείς για μη συμβατικά, συμβατικούς πόρους, πάλι μιλάμε για αέρια του θερμοκηπίου. Αντί λοιπόν να ρίξουμε τόσο βάρος στο συστολιστικό αέριο σε να μην ήταν το σωστό. Το πρόβλημα είναι καινοτομία, αποδοτικότητα των πηγών της ενέργειας, πρωτοποριακός ρόλος που είναι και τα κλειδιά της ανταγωνιστικότητας. Η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και όχι η προσπάθεια ανταγωνισμού στις τιμές. Σε ό,τι αφορά το ρόλο της ανταγωνιστής ε, αποδοτικότητας της, αποδοτικότητας της ενέργειας, πάντα μιλώ εγώ για την ενεργειακή τριάδα η φτηνότερη ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν θα παραχθεί καν. Τα μισά ξοδεύετε για να εξοικονομήσετε μια κιλοβατόρα από ό,τι για να την παραγάγετε. Όταν λοιπόν θα αναπτύξετε την ενιαία αγορά, πράγματι χρειάζεστε την αποδοτικότητα της ενέργειας ως αφετηρία. Και βέβαια και ανανεώσιμες ενέργειες που πάνε χέρι με χέρι μείωση της ενέργειας που καταναλώνετε, που αυτό είναι που χρειάζεται να κάνετε πριν να αναπτύξετε την προμήθεια, την προσφορά. Πόση ενέργεια θα σας χρειαστεί για να περάσει τη μεταβατική περίοδο. Πολύ σημαντικό είναι ο καταναλωτής να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις αβεβαιότητες και με ενδιάμεσα μέτρα. Αποθήκευση για παράδειγμα. Αυτά όλα συνεργάζονται για να ολοκληρώσουν την ενιαία αγορά. Εκεί το κλειδί είναι η αποδοτικότητα της ενέργειας. Όπως είπαμε και το πρωί, δεν χρειάζεται μόνο διασυνδέσεις. Χρειάζεται και τοπική παραγωγή και διανομή. Χρειάζεται συνδυασμός και των δύο και υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτό. Τα ακίνητα επίσης είναι σημαντικό τμήμα της εξίσωσης αυτής, διότι τα ακίνητα απορροφούν 40 περίπου 100 του συνόλου της ενέργειας που καταναλώνουμε. Είναι σημαντικό τμήμα της υποδομής και είναι το ίδιο σημαντικό όπως η δημιουργία και ανάπτυξη των δικτύων. Η τυποποίηση είναι επίση προπόθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και ιδιαίτερα σημαντική για την αποδοτικότητα. Για μένα είναι προϋπόθεση. Αν έχετε τώρα ελάχιστες απαιτήσει για την αποδοτικότητα, eco-design, το σήμα EC, όλα αυτά είναι απαραίτητα για να εναρμοστεί η ενιαία αγορά. Και για τις ανανεώσιμε χρειάζεται κάποια τυποποίηση. Επίσης θέματα ασφάλειας, θέματα πυρασφάλειας των υλικών, όλα αυτά. Εκεί χρειάζεται η εναρμόνιση των, των προτύπων, η τυποποίηση. Πολλά από αυτά ε, υιοθετούνται και παγκοσμίως. Και οι ΗΠΑ ίδιες αυτή τη στιγμή υιοθετούν κάποια ευρωπαϊκά eco-design και εκείνα το ίδιο αυτές οι ευρωπαϊκές νόρμες, τα EN δηλαδή, πάνε να γίνουν τώρα ISO, παγκόσμια πρότυπα. Αν λοιπόν παραγάγετε τώρα πρότυπα για προϊόντα, θα σας επιτρέψουν, να τα θα σας επιτρέψουν αυτά να τα εξαγάγετε, γιατί έχετε αρκετά τυποποιημένα προϊόντα. Και αυτό βοηθεί στις εξαγωγές σας. Επίσης, τα συστήματα ελέγχων της κατανάλωσης ενέργειας, που είναι τμήματα της πρόσφατης νομοθεσίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα, οι έλεγχοι που απαιτούν οι μεγάλες επιχειρήσεις να καθίσουν να εξετάσουν την κατανάλωση ενέργειας, να γνωρίζουν ακριβώς πώς μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειάς τους. Και αυτό λοιπόν είναι σημαντικό κλειδί. Και τα συστήματα διαχείρισης της ενέργειας από τις επιχειρήσεις. Σημαντικό και αυτό. Πολύ δουλειά μένει ακόμα να γίνει στην τελική μορφή και στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς για την αποδοτικότητα της ενέργειας, για την κατάργηση των φραγμών, για την μείωση των δεσποζουσών θέσεων, για οικονομίες κλίμακος, για την αύξηση του εμπορίου, τη μείωση του κόστους, αμοιβαία αναγνώριση επίσης και πιστοποίηση είναι επίσης σημαντικό τμήμα της αγοράς αυτής, της ενιαίας αγοράς δηλαδή. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα αποτελέσει κλειδί και εδώ. Οι βέλτιστες πρακτικές, η έρευνα και ανάπτυξη, η ανταλλαγή πληροφοριών, η συνεργασία. Άλλο πράγμα από την συμπεγνία. Γιατί εκεί υπάρχει αυτή η ισορροπία ανάμεσα στους ε, παίκτες. Επίσης σημαντικό είναι το μακροπρόθεσμο ρυθμιστικό πλαίσιο Χρειάζεται μακροπρόθεσμους στόχους. Επανέρχομαι στους δεσμευτικούς στόχους. Μεγάλη συζήτηση τώρα. Τα περισσότερα από αυτά που βλέπω είναι ότι στόχος ναι, αλλά πρέπει να είναι στόχος αποδοτικότητας. Μόνο στόχος μείωσης δεν αρκεί, γιατί θα υπάρξουν μη οικονομικοί φραγμοί που θα αποτρέψουν την υλοποίησή του. θα πρέπει να είναι στόχοι οι οποίοι να επιτρέψουν και συμμόρφωση με τους στόχους της μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Χρειαζόμαστε ευελιξία λοιπόν. Αυτή θα αποδώσει τα μέγιστα. Λίγα τώρα για, τα, για τις δυνατότητες εξοικονομήσεων. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το δυναμικό εξοικονόμησης σε όλους τους τομείς είναι πάρα πολύ μεγάλο 40% το λιγότερο μέχρι το 2003. 61 για παράδειγμα για τα σπίτια, 26 στη βιομηχανία, 40 και περισσότερο στις μεταφορές. Μεγάλα νούμερα λοιπόν για τα κτίρια όπως είπα που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό σας μίλησα ήδη. Για το 2080 80% δυνατότητα μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτά είναι αποδειγμένα νούμερα από πολύ προσεκτικά διατυπωμένες μελέτες. Εάν οι οικοδομές στην Ευρώπη μπορούν, αν δηλαδή ο ρυθμός ανανέωσής του μπορεί να φτάσει στο 3%, και σε βάθος ανακαινήσεις μπορούν να μειώσουν την ε, κατανάλωση ενέργειας πέντε φορές. Εδώ βλέπετε τα πολλαπλά ωφελήματα της ε, καλύτερης χρήσης της ενέργειας, της πιο αποδοτικής χρήσης της ενέργειας, να μην περάσουμε όλα τώρα. Προσπαθείτε να δείτε αυτό το διάγραμμα που δείχνω τώρα Μπορώ να σας πάρω για παράδειγμα το διαθέσιμο εισόδημα. Η αποδοτικότητα σας δίνει απόδοση της επένδυσής σας. Cash flow επομένως που μπορείτε τις ροές αυτές να τις επενδύσετε αλλού. Μειώνει τη φτώχεια. Βελτιώνει την κοινωνική ευημερία. Δημιουργεί δουλειές. Μισό εκατομμύρια δουλειές μπορούν να φτιαχτούν μέχρι το 2020 εάν συνεχιστεί αυτή η μείωση της ε, χρήσης της ενέργειας, αν αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας δηλαδή συνεχιστεί. Οπότε θα μειωθούν και άλλα, θα μειωθούν οι δαπάνες για την ασφάλιση κατά της ανεργίας και ούτω καθεξής. Βλέπετε ότι η αποδοτικότητα στη χρήση της ενέργειας έχει πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει και χρειάζεται να της δώσει κανείς πολύ μεγαλύτερη σημασία. Ιστορικά, η εξοικονόμηση της ενέργειας είναι το πρώτο καύσιμό μας μεταφορικά. Από εδώ, από, τον, από το γράφημα αυτό της IAA, βλέπετε ότι αν δεν είχαμε χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα μείωσης της ε, κατανάλωσης ενέργειας, η κατανάλωσή μας τώρα πετρελαιοδών θα ήταν 60% περισσότερη από σήμερα. Η αποδοτικότητα της ενέργειας λοιπόν είναι το πιο σημαντικό μας καύσιμο. Και αυτό βασίζεται σε νούμερα και στοιχεία. Πρέπει να ξαναδούμε τα νούμερα αυτά, πρέπει να τα εξετάσουμε πιο προσεκτικά, γιατί είναι πραγματικά εκπληκτικά. Αλλά συγκεκριμένα παραδείγματα. Η Δανία, για παράδειγμα, που έχει αποδείξει, έχει υψηλούς φόρους κατανάλωση ενέργειας και όμως είναι από τι πιο ισχυρέ οικονομίε στην Ένωση. Άρα το επιχείρημα ότι οι φόροι καταστρέφουν τη βιομηχανία δεν είναι αληθεία. Και αυτά τα δείχνει πρόσφατη μελέτη στη Δανία. Δεν έχουν σχεδόν καμία επίπτωση στον ιδιωτικό τομέα, στην απασχόληση ή στην κατανάλωση ή στο ισοζύγιο πληρωμών όλα αυτά που έχουν θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή στην απασχόληση. Δημιούργησε και έναν μεγάλο αριθμό ε, επιχειρήσεων καθαρής τεχνολογίας. 10% του ΑΕΠ της, παρόλο που είναι μικρή χώρα, είναι από τις, έχει από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις όπως Danfoss, Vestas, Grundfos, Rohul, Siemens, Velux και πολλές ε, εταιρείε χορήγησης συμβουλών, παροχή συμβουλών. Και το 10% της συνολικής, των συνολικών μάλλον δανέζικων εξαγωγών είναι προϊόντα τέτοια καθαρής τεχνολογίας. Βλέπετε εδώ νούμερα που, βλέπετε, που δείχνουν ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία επίπτωση στους παράγοντες του ΑΕΠ. Αντί θέτα μάλιστα αυξάνει την απασχόληση. Η Δανία κάτω-κάτω είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θετικό απολογισμό στην ενέργεια. Και η Μάλτα πάνω πάνω 100% εξαρτώμενη από τις εισαγωγές ενέργειας. Είναι λοιπόν πραγματικά εντυπωσιακά τα νούμερα αυτά και έχουν σχέση και με τον τρόπο που χειρίζονται οι Δανείοι την ενέργειά τους. Εδώ τώρα λίγα στοιχεία για το δυναμικό εξοικονόμησης Ε, χώρες όπου έχουν χρησιμοποιήσει το CHP και την ανάκτηση της θερμικής ενέργειας μεταξύ 20 και 30%. Το ίδιο για τις τσιμεντοβιομηχανίες. Πολύ ψηλό βλέπουμε από τα, ΟΣΑ, από τα στοιχεία του ΟΣΑ τις δυνατότητες εξοικονόμησης και για το CHP και για την ε, ανάκτηση θερμικής ενέργειας. Το ίδιο για τα χημικά. Υπάρχει η ικανότητα λοιπόν της βιομηχανίας για εξοικονόμηση. Αυτά είναι τα νούμερα που είπε προηγουμένως η Business Europe. Η μείωση των τιμών της ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτά θα διαρκέσουν για πάντα. Εν τέλει, η ενιαία αγορά πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με επενδύσεις, πρέπει να εξετάσει όμως την εξοικονόμηση ενέργειας, πρέπει να βασιστεί στις ανανεώσιμες οι δουλειές που θα προέλθουν από τον πράσινο άνθρακα είναι ε, αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη ασφάλεια, θα πρέπει να γίνουμε πρωτοπόροι και να έχουμε και στόχους εξοικονόμησης. Τώρα τέλος μια μικρή εικόνα που με εντυπωσίασε πολύ ίσως να την έχετε δει. Είναι ο δορυφόρος Τζούνο που στάλθηκε στον Δία. Χρησιμοποιώντας ε, πολύ ε, πρωτόγονη ε, τεχνολογία για τα σημερινά μάτια. Την έκανα να κάνει μερικές βόλτες γύρω από τη γη για να πάρει φόρα και μετά εκτοξεύθηκε να πάει προς τον Δία και τώρα έχει μπει σε τροχιά γύρω από τον Δία. Για πρώτη φορά. Αυτή τη γη που την που ζούμε σε αυτήν τόσα εκατομμύρια χρόνια, πρώτον δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας στο διάστημα, δεύτερον η τεχνολογία μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα και μπορεί να λύσει και το πρόβλημα των τιμών στο οποίο έχουμε κολλήσει τώρα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, κύριε Μπόι, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για, τις, ε, για την ενεργειακή απόδοση. Είμαστε λίγο πίσω στο πρόγραμμα, αλλά δεν διέκοψε κανένα γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσε όλε οι εισηγήσει. Υπενθυμίζω σε όλου ότι όσοι θέλουν να μιλήσουν και από εθνικά κοινοβούλια πρέπει να συμπληρώσουν το κόκκινο χαρτάκι. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι όπως και το πρωί. Δύο λεπτά για τον κάθε ομιλητή και ένα λεπτό για τις ερωτήσεις. Δύο ομιλητές λοιπόν από τα Εθνικά Κοινοβούλια και ενα από το Ευρωπαϊκό. Ο πρώτος των καταλογών μου των ομιλητών είναι συνάδελφος από το Κωσοπέδιο, το Κόσοβο, την Επιτροπή Οικονομίας και Ανάπτυξης. Είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. σα Ασοκέα. Με συγχωρείτε αν δεν πρόφερα σωστά το όνομά σα. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να πω ότι στο Κόσμο αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένα παραγωγό. Είναι ε, ο μόνος ε, έχουμε ιδιωτικοποιήσει την διανομή ενέργεια επίση. Ετοιμάζουμε νομοθεσία όμως για το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζουμε και νομοθεσία για τις συντηρητικές επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στο κόσμο για μικρής κλίμακας έργα. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε διασύνδεση με την Αλβανία που θα μας δώσει τη δυνατότητα να έρθουμε πιο κοντά σε μια ενιαία αγορά ενέργειας. Επίσης, δρομολογήσαμε το σχέδιο δημιουργίας ενός νέου σταθμού παραγωγής ενέργειας ε, και έχω σαφώς δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά τις επιδοτήσεις για τις ανανεώσιμες. Μάλιστα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κ. Μπέγερ σχετικά με τις επιχειρήσεις του τομέα. Ποια είναι τα ωφελήματα από τις επιδοτήσεις και πώς επηρεάζουν την αγορά και τις επιχειρήσεις. Ο κ. Μπέγερ επίσης ανέφερε την μείωση των εκπομπών. επηρεάζει αυτό επιθετικά, αν επηρεάζει τις επιχειρήσεις και πώς βλέπουν οι επιχειρήσεις τον ρόλο τους προκειμένου. Τις ωφελεί η μείωση των εκπομπών και τι γίνεται με τις επιδοτήσεις, όπως προείπα. Και πόσο καιρό θα χρειαστούμε επιδοτήσεις. Σάλφη να είμαστε πιο σύντομοι γιατί δεν θα μιλήσουν όλοι όσοι θέλουν. Παρακαλώ και θα πρέπει να σας διακόπτω εγώ και δεν θέλω. Λοιπόν, άλλη μια ερώτηση όσον αφορά τις διαφάνειες που είδαμε. Επειδή κάποιος το έθεσε, θα σας στείλουμε, μπορούμε να σας στείλουμε την παρουσίαση μέσω email στις διευθύνσεις σας. Από την πολιτική ουσία, Στανισλαβ Ιβάν. Ε, σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είδατε τους τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής ενέργειας. Εγώ πιστεύω ότι μόνο μια πολιτική συνοχή μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάπτυξης στην Ευρώπη. Δεσμευόμαστε φυσικά, αυτό δεσμευόμαστε για μείωση των εκπομπών, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μπούμεραν για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. αυτά συνδέονται και με την πολιτική για το κλίμα. Το αποτέλεσμα είναι όμως υψηλές τιμές για την ενέργεια. Αυτό αποτελεί πρόσκομα στην ανάπτυξη. Δείτε στην την Πολωνία. Και μια μικρή αύξηση λίγων ποσοστιαίων μονάδων στην τιμή της ενέργειας θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Αυτό είναι μείζον κίνδυνος. Και έχουμε και την λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής δικαιωμάτων εκπομπών. Πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε την αγορά λοιπόν να κάνει τη δουλειά της. Να ευχαριστήσω επίσης την προσοχή σας στο γεγονός ότι πρέπει η Ευρώπη να επιστρέψει στον δρόμο της ανάπτυξης. Η τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών δεν είναι δυνατόν να επηρεάζει την τιμή της ενέργειας. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τις δημορφίες του ενός ή του αλλού κρατούς μέλους, την γεωγραφική θέση, καταρχήν, μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σύμπασας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συναδελφοί, μιλούμε για την αποδορική χρήση της ενέργειας. Ξέρουμε ποιος είναι ο βασικός μας στόχος για το 2030. Βλέπουμε τώρα τα στατιστικά στοιχεία. Βλέπουμε πώς αυξήθηκε η κατανάλωση από το 8 στο 2012. Ελπίζουμε παρόλα αυτά να πετύχουμε τους στόχους μας. Η αποδορική χρήση της ενέργειας προϋποθέτει την, τον εξυγχρονισμό των κατοικιών, κατά το οποίο αφορά ακόμη περισσότερο την Ανατολική Ευρώπη. Εδώ υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας. Όσον αφορά τώρα τις ανανεώσιμες. Πώς θα ενταθεί η χρήση τους. Πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες οι οποίοι θα αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες τα σπίτια τους. Το είπαν πολλοί ομιλητέ. Είπαν ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε τη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Ωραία, υπάρχει όμω κάτι, επαναλαμβάνω, για τα νοικοκυριά και τη χρήση των ανανεώσιμων στα νοικοκυριά. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Ο λόγος τώρα σε έναν Έλληνα συνάδελφο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ανάγκη για μια ενεργειακή πολιτική που θα ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και τα σημαντικότερα βήματα για να επιτευχθεί αυτό ο στόχο είναι τα παρακάτω. Πρώτα απ' όλα η αξιοποίηση του υφιστάμενου πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση που κατευθύνει τι πολιτικέ τη για την ενέργεια και το κλίμα στο 2020. Συγκεκριμένα, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, η υποστήριξη τη ανάπτυξη ανταγωνιστικότητα και των θέσεων εργασία μέσα από την εφαρμογή προσέγγιση που αποτελεί συνδυασμό υψηλή τεχνολογία αποδοτικότητα σε θέματα κόστου και αποδοτική χρήσης πόρων. Σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, οι πολιτικέ για την ενέργεια και το κλίμα μπορεί να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για τη ζήτηση και την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρο στο τομέα των καθαρών και ενεργειακών αποδοτικότερων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών και των οικολογικών τεχνολογιών. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Πολλέ από τι πολιτικέ αυτέ συμβάλλουν επιπλέον στη μείωση τη ατμοσφαιρική ρήπανση και στη βελτίωση τη υγεία. Παράλληλα, οι πολιτικέ έχουν επικριθεί επειδή ασκούν αρνητική επίδραση στι τιμέ τη ενέργεια και επηρεάζουν αρνητικά τον οικονομικά προσιτό χαρακτήρα τη ενέργεια για τα νοικοκυριά και την ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων κλάδων. Γι' αυτό έχει σημασία να φροντίσουμε για την πλήρη εφαρμογή τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά Επίση, είναι αναγκαίο να καταστεί δυνατή η μελλοντική εκμετάλλευση των εγχώριων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, τόσο από συμβατικέ όσο και από μη συμβατικέ πηγέ, με περιβαλλοντολογικά ασφαλή τρόπο. Τέλο, χρειάζεται διαφοροποίηση των οδών ενεργειακού εφοδιασμού, που να μπορεί να βελτιώσει τον ανταγωνισμό στι αγορέ ενέργεια, ενώ θα μπορούσε να επιτευχθεί σημαντική μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση από επενδύσει σε ενεργειακή απόδοση όπω σε κατοικίε η περαιτέρω εμπόδιση, εμπέδωση τη ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και μεταφέροντα την εμπειρία από τη χώρα μου με πλούσιου ανταγωνιστικού πόρου αλλά μικρή συγκριτική εκμετάλλευση, πρέπει να συνοδεύεται από βελτίωση τη διαχείριση των διασυνδεμένων δικτύων, μείωση του κόστου και βελτίωση των επιδόσεων των τεχνολογιών, καθώ και από συνεχή στήριξη καινοτομία. Ευχαριστώ. E, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάλστης από το Λιθουανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Θέλω να απευθυνθώ στον εκπρόσωπο του Business Europe ε, γιατί δεν ε, οθείτε τις εταιρείες σας να αλλάξουν από την καφέ στην πράσινη οικονομία αν είστε αρκετά υπεύθυνο, θα πρέπει να κάνετε ένα σχεδιασμό για την ανάπτυξη των επιχειρησιών σα για τα 10-20 επόμενα χρόνια. Και πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι η διαγωνιστικότητα τη οικονομία σε 10 χρόνια θα προσμετράται από την αποτελεσματικότητα των ενεργειακών χρηστών και η υποδοτικότητα σημαίνει και μεγαλύτερο κέρδος για τη βιομηχανία και συμμόρφωση με τους στόχους κλιματικής αλλαγή και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, είναι το ε, η απάντηση, όχι το σχιστολιθικό αέρια, όχι τα καταστροφικά πυρηνικά, ούτε η δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα με τις ενώσιμες πηγές ενέργειας ε, να μειώνονται ως προς το κόστος ε, κάθε χρόνο σε 10 χρόνια θα είναι πιο ανταγωνιστικές και χωρίς επιδοτήσεις και αυτό δεν ισχύει για την πυρηνική ασφαλεία του σχιστολιθικού αέριο η Business Euro μίλησε με τη Σεύρον για να, να μιλήσει στην Σεύρον για να επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι στο στελθικό αέριο και να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υιοθετηθεί νομοθεσία για να ανοίξουν τα ευφυή δίκτυα στην Ευρώπη. Μόνο τότε όσα κάνετε θα είναι βιώσιμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Πρόντι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να αναφερθώ στα όσα είπε ο κ. Πρόκ σε σχέση με την ηλεκτρική ενέργεια και την αναγκαιότητα να έχουμε είτε συσσόρευση ενέργειας αλλά και συσσόρευση θερμότητας. Και θα ήθελα να πω ότι η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την υπερπαραγωγή ενέργειας για να παράξουμε υδρογόνο και επομένως ε, να εφοδιάσουμε τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν απευθείας υδρογόνο όπως τα δηληστήρια, ε, οι βιομηχανίες λιπασμάτων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να συνεισφέρουμε στην ισορροπία του ηλεκτρικού δικτύου και ταυτόχρονα να προσέξουμε και σε άλλες τεχνικές αποθεματικού. Και παραδείγματο χάρη με στην ε, παραγωγή ολικής ενέργειας σε υπεράκτες πλατφόρμες ε, θα μπορούσαμε να μετακινήσουμε έναν όγκο υδάτων που βρίσκονται κάτω από αυτές τις πλατφόρμες έτσι ώστε να αποτελούν ε, το απόθεμα, απόθεμα για αυτές τις εγκαταστάσεις της υπεράκτειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, πάντως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Τσίρου από το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπόθηκε εδώ ότι στην Αμερική υπάρχει πιο φτηνή και πιο καθαρή ενέργεια και συμφωνούμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα και πιστεύω ότι οι κύριες προκλήσεις ε, που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη είναι να έχει καθαρή ενέργεια σε πιο φτηνές τιμές. Παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον ε, την ε, παρουσίαση του κυρίου Μπάουι. Μας είπε ότι αυτό που έχει σημασία δεν είναι η τιμή αλλά το κόστος. Θέλω να κάνω μια ερώτηση κύριε Μπάουι. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενθαρρύνει σχέδια για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χωρίς να έχει ένα κοινό σύστημα για το ενεργειακό μείγμα για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. που θα μπορούσε να διασφαλίσει το ίδιο κόστος ε, των υπηρεσιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το σύστημα υπολογισμού για την ενέργεια που θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών μελών θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρώτη λύση για να λύσουμε το πρόβλημα του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Σχεδίου. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπρίτε από το Λιθωνικό Κοινοβούλιο. Κυρία Λέτου η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι στενά συνδεδεμένη με την ενιαία αγορά ενέργειας. Αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε λοιπόν από την Κομισιόν είναι να διαχωρίσει τις τιμές του πετρελαίου από τις τιμές του φυσικού αερίου και να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική αγορά αερίου. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τους ομιλητές σε σχέση με την ενεργειακή εξοικονόμηση και την ενεργειακή αποδοτικότητα στην ε, κατασκευαστική βιομηχανία, στα κτίρια και στις μεταφορές. Γιατί πράγματι αυτό το καθήκον πρέπει να επιτελέσουμε. Υποτίθεται ότι ο 21ος αιώνας θα ήταν ο αιώνας της πράσινης οικονομίας και της πράσινης ενέργειας. Από όσο βλέπω εγώ μέχρι τώρα, δεν ε, είναι αυτός πλέον ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, θα συνιστούσα να δούμε ποιοι είναι οι πρωτοπόροι, να τους παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς, τους πρωτοπόρους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Δανίας και άλλες, Δανία και άλλες χώρες, γιατί αυτή είναι το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κορέρετε Κάμπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τη Λιθωνική Προεδρία και τους συναδελφούς από τα Εθνικά Κοινοβουλία που παρευρίσκονται εδώ. Θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το ότι εμείς ε, οι Ευρωπαίοι τελικά οδηγηθήκαμε σε μία ε, πλάνη, δηλαδή προβήκαμε στην αποβιομηχανοποίηση και τώρα θέλουμε να κάνουμε μία νέα βιομηχάνηση για να μπορέσουμε να αντιγωνιστούμε όχι μόνο με την Κίνα αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι παράδοξο που σε αυτή τη σημερινή συνάντηση ε, υπήρξε μία αντιφατική παρέμβαση και αυτή η συζήτηση είναι αντιφατική. Εμείς ακούσαμε τι γίνεται με το συγχυστολιστικό αέριο και έγινε αναφορά και στη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ε, κλιματικές αλλαγές ε, και τελικά τι πρέπει να κάνουμε, να καταλαβαίνουμε περισσότερο άνθρακα από τις ΗΠΑ γιατί ε, εκεί είναι πιο φθηνός ο άνθρακας, ο άνθρακας που έρχεται από εκεί, από το αέριο που έχουμε εδώ. Τελικά όμως πρέπει εμείς να δούμε ποιες είναι οι ευρωπαϊκές αξίες και να αναπτύξουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα που είναι μια παγκόσμια αξία. Τώρα, η ασφάλεια του εφοδιασμού. Σε ορισμένες χώρες βλέπουν να υπάρχει ένας πολιτικός κίνδυνος για το θέμα αυτό και αυτός ο κίνδυνος πρέπει να μεταφραστεί σε πλεονέκτημα τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας πρέπει να οικοδομηθούν και να καταπολεμήσουμε την ενεργειακή απομόνωση. Η Ευρώπη έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αυτό πρέπει να περασπίσουμε. Τέλος, εγώ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται με τις ανανεώσιμες. Έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ανανεώσιμες και τώρα από ό,τι φαίνεται έχασε τον ενθουσιασμό της. Δεν μπορούμε να χάνουμε τον ενθουσιασμό μας, ε, δεν μπορούμε να σκοτεινιάζει συζήτηση όταν μιλάμε για τα κίνητρα ή όταν μιλάμε για το υπολογισμό του κόστου. Ευχαριστώ. Στον επόμενο, ο είναι ο κύριο Ντέβιτ Κρύπα από το Ιταλικό Κοινοβουλίο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους κύριους Μπλοκιμπάου για τις ε, ομιλίες τους. Νομίζω ότι το σχετικό ε, αέριο αποτελεί παραπλάνηση, μια φθαλμαπάτη ε, Επομένως, η ιστορία της αντιγωνιστικότητας της βιομηχανίας ε, ουσιαστικά θα εκμηδενιστεί ότι ε, όλοι θα ευθυγραμμιστούν στο συστολικό αέριο. Αντίθετα, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα για την τρίτη ε, βιομηχανική επανάσταση, δηλαδή ότι υπάρχει μια προοπτική εξόδου που αναφέρθηκε από τον Τζέρεμι Ρίφκιν. Μια άλλη πτυχή είναι η εποδηπεδετικότητα ε, που αποτελεί ε, ουσιαστικά το κύριο πλεονέκτημά μας. Ε, αυτό είναι ένα πλεονέκτημα και κυρίως για όσους έχουν αναπτύξει κάτι τέτοιο προς αυτήν την κατεύθυνση. Η αποθεματοποίηση, η αποθηκευσή πρέπει να έχει πρωταρχικό ρόλο, όμως... Πρέπει να γίνεται από κοινού με τον καταναλωτή. Ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να διαφοροποιήσει σε ποια φάση, σε ποιο στάδιο θα καταναλώνει η ενέργεια. Δηλαδή πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να διαφοροποιήσει την τιμή κατανάλωσης ε, το βράδυ σε σχέση με τι άλλες ε, ενεργειακές προσφορές έχει. Εμείς στην Ιταλία έχουμε διάφορα στάδια ε, χρονικά διαφοροποίησης των τιμών. Όμως δυστυχώς συμβαίνουν κάποιες συμπεριφορές που τελικά οδηγούν στο να χαθεί ένα τέτοιο πλεονέκτημα. Τι συμπεριφορές δεν μπορούμε να τις επιτρέψουμε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μπεναμάτη από το Ιταλικό Κοινοβούλιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απογευματινή συνεδρίαση ασχολείται με ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα μου, τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε μεγάλη εκτίμηση τα λόγια του κυρίου Ταγιάννη, γιατί θεωρούμε ότι είναι σκόπιμη ιδέα η Ευρώπη να περάσει σε πολιτικές ανάπτυξη μετά από αυτό το στάδιο των πολιτικών περί ε, για μια πολιτική ανάπτυξης και αντιγωνιστικότητας δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς μια ενέργεια με αντιγωνιστική τιμή και κόστος ε, σε παγκόσμιο επίπεδο και που να μπορεί να συγκριθεί στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό το λόγο εγώ θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είπα και το πρωί, στο ρόλο της αγοράς. Ο ρόλος της αγοράς είναι απαραίτητο στο σημείο αυτό και σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό του συστήματος, ε, τις διασυνδέσεις, ε, ε, και ε, την διαχείριση αλλά και από τη σκοπιά της απελευθέρωσης των εσωτερικών αγορών. Μόνο αυτό μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικότητα και να οδηγήσει σε πτώση των τιμών για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Ένα τελευταίο σημείο για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Εμείς θεωρούμε ότι η αποδοτικότητα μεταξύ άλλων θεμάτων, που δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ, η ενεργειακή αποδοτικότητα έχει ένα θεμελιώδη ρόλο για το μέλλον για το σύστημα της παραγωγής αλλά και για το βιομηχανικό σύστημα και σε αυτό το θέμα αλλά και για τις ανανεώσιμες θα πρέπει να δώσουμε μία ενίσχυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε ιδιαίτερα όταν θα προετοιμάζουμε τα νέα προγράμματα. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Τελευταίος, ο η Ευρωβουλευτής Ντεκράτσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. και Καρβάγιο. Απευθύνω χαιρετισμό και στους άλλους ευρωβουλευτές και στους συναδέλφους μου από τις Εθνικές Βουλές. Έχω μια ερώτηση και προς άλλους ομιλητές, αλλά ιδίως στον κύριο Μπόη. Συμφωνώ με την ανάγκη της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας. Ωστόσο, αντί να επικεντρωθούμε μόνο σε αυτό, νομίζω ότι ως policy makers πρέπει να αφήσουμε ανοιχτές όλες τις εναλλακτικές επιλογές, όπως περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη για να μειώσουμε το κόστος των ανανεώσιμων ενεργειών, διότι στο παρελθόν έχουμε κάνει το σφάλμα να επιδείξουμε ορισμένα στάδια της ανάπτυξης των τεχνολογιών αυτών που δεν ήταν ακόμη όριμες. Πρέπει λοιπόν να το κάνουμε αυτό, πρέπει να ολοκληρώσουμε την ενιαία αγορά και πρέπει να αναζητήσουμε και εναλλακτικέ πηγές ενέργειας και να αναζητήσουμε τρόπους να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Να ρίξουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας σε διαφορετικές τεχνολογίες γιατί για την περίπτωση της Ευρώπης που έχει πολλές ιδιαιτερότητες δεν έχουμε δηλαδή τεράστιους πόρους ενέργειας μόνο εάν ενώσουμε όλες τις προσπάθειες αυτές μπορούμε να φτάσουμε σε καθαρή φθηνή και διαθέσιμη ενέργεια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους, λέει ο Προεδρεύων και ο Ζεμαϊτάιτης. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις και άλλα σχόλια και τώρα θα δώσω τρία λεπτά στους ομιλητές για να μπορέσουν να απαντήσουν. Με πρώτον κύριο Μπέιρερ από την Ένωση Business Europe. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλες τις παρεμβάσεις σας που πραγματικά είναι πολύ τιμές. Έγιναν πολλά σχόλια στα οποία θα ήθελα να επανέλθω. Είναι λίγο δύσκολο να το κάνω γιατί έχω έξι σελίδες σημειώσεις. Θα προσπαθήσω ωστόσο να αναφερθώ στα πιο σημαντικά. Και ευρωβουλευτές και εθνικοί βουλευτές αναφέρθηκαν στην διασύνδεση στην ενιαία αγορά. Βεβαίως, αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε όλοι είναι να φτάσουμε σε φθηνές τιμές ενέργειας και κόστος και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να προωθήσουμε τους στόχους μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προωθήσουμε την ενιαία αγορά, άρα περισσότερο ανταγωνισμό και αυτό σημαίνει βέβαια διασύνδεση. Γνωρίζω ότι τα συζητούμε αυτά εδώ και πολύ καιρό, είναι και θέμα και στην Λιθουανία, σημαντικό θέμα, αλλά και στην Ιβυρική Χερσόνησο. Για τις επιδοτήσεις. Ποιε είναι οι επιπτώσεις στις εταιρείε. Βεβαίως, αν έχετε μια αναλογία 11% σε ένα project, τότε αυτό είναι βέβαια ο στόχος των επιδοτήσεων όταν μιλούμε για ανανεώσιμες ενέργειες. Όπως είπα, είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων ενεργειών. Δεν είμαστε όμως υπέρ διαρκών μόνιμων επιδοτήσεων και μόνιμων μεταφορών. Ιδίως όταν αυξάνουν το κόστος, στρεβλώνουν το ε, σήμα για τις εκπομπές διευθυντών του άνθρακος. Σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα ενέργειας, να μην παρανοηθώ, συμφωνώ με τα όσα είπαν πολλοί από τους άλλους. Πολλές επιχειρήσεις κάνουν σημαντική προσπάθεια εξοικονόμηση τη ενέργειας και επενδύοντας πολλά γιατί συχνά είναι και ο πιο οικονομικός τρόπος να μειώσει κανείς τις ανάγκες του σε ενέργεια. Από την άλλη μεριά δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε ιδιαίτερο στόχο γι' αυτό. Χρειαζόμαστε ένα συνολικό σύστημα το οποίο θα αφήσει στην αγορά τη δυνατότητα να καταλήξει στις πιο αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις για τις καθαρές τεχνολογίες. Πάλι εδώ, μην με παρανοήσετε. Αυτό, όχι όμως, αυτό είναι όχι μόνο το μέλλον, είναι και το παρόν και των δικών μας μελών. Και το υποστηρίζουμε και πολύ. Και είμαστε υπέρ της μεταλλαγής της ευρωπαϊκής οικονομίας σε low carbon economy. Πρέπει να το κάνουμε όμως με κάποιο ρυθμό και με κάποιο κόστος που θα επιτρέψει στην πλειοψηφία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να παραμείνει ανταγωνιστική. Και όπως είπε ο συνάδελφός σας από την Πορτογαλία στο τέλος, βεβαίως και πρόκειται για την σύγκριση σε παγκόσμιο επίπεδο. Και στην σύγκριση σε παγκόσμιο επίπεδο βλέπουμε ότι χάνουμε ανταγωνιστικότητα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Δυο ακόμη σχόλια ή ένα αν θέλετε. Μια στιγμή παρακαλώ. Για το σχιστολιθικό αέριο. Δεν θέλω να πω σε πολλές λεπτομέρειες για το σχιστολιθικό αέριο. Γνωρίζουμε ότι από μόνο του δεν θα λύσει όλα μας τα προβλήματα. Θα πρέπει όμως να συναποτελέσει τμήμα του energy mix και πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση βασισμένη στις πραγματικές ενδείξεις. Εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε τους κινδύνους. Δεν λέμε ότι πρέπει να γίνει εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου με οποιοδήποτε τίμημα πρέπει να συζητήσουμε απαλλαγμένοι από ιδεολογίες, από μύθους και βασισμένοι σε πραγματικά στοιχεία. Αυτό το χρωστάμε και στις, και οικονομίες και στους λαούς της Ευρώπης, γιατί νομίζουμε ότι είναι η σωστή προσέγγιση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον καθηγητή κύριο Μπλοκ του Πανεπιστημίου τη Ουτρέχτης. Ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Ώρες ολόκληρες θα μπορούσαμε να συζητούμε τα θέματα αυτά, αλλά εγώ θα έρθω σε ορισμένα σχόλια. Πρώτα, πώς μπορούν οι ανανεώσιμες ενέργειες να δώσουν όθηση στις επιχείρησεις. Μπορούν. Το καλύτερο παράδειγμα είναι πάλι η Γερμανία, όπου βλέπουμε να ανθούν οι βιομηχανίες ανανεώσιμης ενέργειας με χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης, έστω και αν έχουν χάσει ένα μερίδιο της αγοράς από την Κίνα, που πήγε στην Κίνα δηλαδή, παραγωγή κινέζικη. Όμως το μεγάλο μέρος έντασης εργασίας αλλά και έντασης αξίας βρίσκεται στη Γερμανία και θα προσφέρει νέες δυνατότητες, νέα απασχόληση και όθηση. Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε από πλευρά σας είναι πώς μπορούν να οθηθούν τα νοικοκυριά να επενδύσουν στην ανανεώσιμη ενέργεια. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Διάφορες χώρες κάνουν διαφορετικά πράγματα στη Γερμανία έχουν το feed-in, την διοχέτευση δηλαδή στα δίκτυα και φθηνά δάνεια διότι βεβαίως δεν έχει το κάθε νοικοκυριό τις απαραίτητες καταθέσει στην τράπεζα για να μπορέσει να κάνει τη σχετική επένδυση αλλού χρησιμοποιούνται άλλα συστήματα καμιά φορά είναι επικίνδυνο διότι δεν μπορεί να διατηρηθούν για μακρόχρονικό διάστημα Υπάρχουν λοιπόν διάφορες επιλογές, υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Ο Δόκτωρ Πρόντι έκανε την ερώτηση αν θα πρέπει ίσως να μετατρέψουμε το υπερβάλλον ηλεκτρικό ρεύμα σε υδρογόνο. Αυτό βέβαια δεν είναι βραχυπρόθεσμη λύση. Το ζήτημα είναι ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι σημαντικός φορέας ενέργειας και πολλοί πολύτιμότερο από οποιονδήποτε άλλο. Όσο μπορεί να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρικό ρεύμα, καλύτερα να το χρησιμοποιείς, καλύτερα να το χρησιμοποιήσει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά ω ηλεκτρικό ρεύμα παρά να το μετατρέψει επιτόπου σε υδρογόνο. Και η τελική ερώτηση είναι, γιατί χάνουμε τον ενθουσιασμό μα σιγά σιγά για τι ανανεώσιμε ενέργειες, μία από τι ερωτήσει που τέθηκε. Νομίζω ότι πολλοί εξακολουθούν και είναι ενθουσιώδει οπαδοί τη ανανεώσιμη ενέργεια και κυβερνήσει βλέπουμε ότι περνούμε τώρα σε μια κατάσταση όπου οι ανανεώσιμες ενέργειες ήταν, είχαν περιορισμένο μερίδιο. Βλέπουμε τώρα τις μεγάλες συνέπειες. Μιλάμε πλέον για γίγαβατ παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και βέβαια προχωρούμε σε διαφορετικές καταστάσεις. Βλέπουμε επίσης και τα καλά αποτελέσματα μειώσεις των εκπομπών, καλύτερες τιμές Βλέπουμε την απασχόληση που παράγεται. Βεβαίω υπάρχουν προβλήματα που μπορούν όμως να επιληθούν. Αυτή λοιπόν είναι, τώρα είναι λοιπόν η ώρα, η κρίσιμη στιγμή. Κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε τι γίνεται και μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό και να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας ο λόγος στον Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενεργειακά αποδοτική οικονομία, κύριε Πάουε. Πολύ σύντομα, ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις, πολύ χρήσιμες. Ένα σχόλιο σχετικά με το πώς οι επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση επηρεάζουν το κόστος της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι προκειμένο ότι υπάρχει φόβος για επενδύσεις το οποίο αφορά επενδύσεις παντού στην παραγωγή ενέργεια, στα δίκτυα κλπ. Εδώ οι επενδύσεις είναι μακροπρόθεσμες. Πρέπει λοιπόν ο υπολογισμός να αφορά όπως τα κτίρια, τη διάρκεια, τη συνολική διάρκεια ζωής ενός κτίριου, 30, 40, 50 χρόνια και περισσότερο και μετά να γίνει μια υφαίρεση και αναγωγή στην καθαρή παρούσα αξία και έτσι να συνεκτιμηθούν οι χρηματικές ροές. Διότι η επένδυση εδώ σημαίνει ότι μειώνω την κατανάλωση ενέργειας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πληρώνω λιγότερα για ενέργεια. Λοιπόν, θα πάρει λίγο χρόνο αυτή η υπόθεση, αλλά είναι βέβαιο ότι η καθαρή παρούσα αξία είναι σαφώς θετική. Οι υπολογισμοί ποικίλουν βεβαίω, αλλά γενικά δεν υπάρχει καμία φωλία για το συμπέρασμα αυτό. Όσον αφορά τις ανανεώσιμες, υπάρχει και μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή. Είναι η λεγόμενη καμπύλη μάθησης. Όταν κάνεις επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, για παράδειγμα, πέρα από την έρευνα και την ανάπτυξη, υπάρχει και μάθηση μια σταδιακή εξοικείωση. Μαθαίνεις πώς να επιτυγχάνεις εξοικονόμηση ενέργεια με πιο φθηνό τρόπο. Άρα το μοναδιαίο κόστος πέφτει και αυτό με το χρόνο. Όλο και περισσότερο μάλιστα. Συμφωνώ επίση απολύτως για την έρευνα και την ανάπτυξη. Πρέπει να είσαι μπροστά. Η πράσινη τεχνολογία και αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς τελειώσαμε με την έρευνα και την ανάπτυξη. Και τέλος, όσον αφορά τους στόχους. Οι στόχοι στην απόδοση ή στο ποσοστό των ανανεωσίμων είναι, ξέρετε, και ένα εργαλείο ρύθμισης της αγοράς. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, μάλιστα, να πειράσει την αγορά Γι' αυτό τα κρατημέλη πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αξιόπιστα ποιοτικά στοιχεία. Να θέτουν στόχους και μετά να αφήνουν την αγορά να αντιδράσει. Κάνε το όπως θέλετε από εκεί πέρα. Αυτός είναι ο στόχος. Προσαρμόζοντας την προσπάθεια στις τοπικές ανάγκες, δημορφίε κλπ. Δώστε ευελιξία. Και αυτό είναι και η ομορφιά, αν θέλετε, ενό στόχου. Ότι θέτει το στόχο και φέρνει τους άλλους μετά να το πετύχουν όπως κρίνουν πιο πρόσφορο. Αυτό ισχύει και τις ανανεώσιμες και το σχετικό στόχο. Οι επενδυτέ, η αγορά, η βιομηχανία θα βρουν τον δρόμο τους εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Γιατί όλοι αυτοί χρειάζονται χρόνο να σχεδιάσουν, να επενδύσουν. Μια βιομηχανία δεν παράγει ξαφνικά καλύτερα μονοτικά, είναι μία νυχτή. Όλοι αυτοί χρειάζονται μακροπρόθεσμους στόχους και μεγάλες προθεσμίες. Τότε και μόνο θα επενδύσουν και τότε θα έχουμε ανάπτυξη, νέες θέσεις απασχόλησης και όλα τα ωφέλη για την κοινωνία που προέρχονται από τις επενδύσεις, από την υψηλότερη απόδοση και την αυξημένη χρήση ανανεωσίμων πλέον ενέργειας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Από τη συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα, φτάνουμε προς το τέλος. Ας κλείσουμε τη σημερινή συζήτηση. Θέλω λοιπόν στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω ειλικρινά την Επιτροπή Ήτρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την κυρία Σαρτόρη, την Πρόεδρο και την Αντιπρόεδρο, την κυρία Τόγια η οποία με βοήθησε ως ε, συμπρόεδρο τη απογευματινή συνεδρία. Να ευχαριστήσω επίση για αυτήν την ευκαιρία συνδιοργάνωσης μιας πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησης. τη συνάδελφη. να ευχαριστήσω τους ομιλητές. Ακούσαμε διάφορες απόψεις. Συζητήσαμε με τη συμμετοχή και βουλευτών από από εθνικά κοινοβούλια να υπογραμμίσω ότι μια αποδοτική αγορά ενέργειας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς διασυνδέσεις. Αυτό το υπογραμμίσαμε και σήμερα. Οι ομιλητές επίσης ανέφεραν α, τις λεγόμενες ενεργειακές νησίδες, περιοχές αποκομμένες από το υπόλοιπο δίκτυο. Υπό Λιθουανική Προεδρία καταφέραμε να εγκρίνουμε έναν κατάλογο 248 PCI για να μπορέσουμε να ενοποιήσουμε την αγορά και να αποφύγουμε τις ενεργειακές νησίδες. Συνάδελφοι, ο στόχος μας είναι η υψηλότερη απόδοση στη χρήση της ενέργειας. Έχουμε ένα πρόγραμμα, ο πρόεδρος, η πρόεδρος είπε ότι χρειαζόμαστε και κανόνες και επικοινωνία. Αυτό είναι σημαντικό τόσο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία όσο και για τα νοικοκυριά. Η ανταγωνιστικότητα, ευκαιρίες αξιοποίηση των πόρων διασυνοριακά σημαίνουν μεταξύ άλλων καλύτερε μέρε και για τι μικρομεσαίε και άλλε επιχειρήσει. Το σημερινό σύστημα ευνοεί μάλλον τι μεγάλε επιχειρήσει. Οι μικρομεσαίε θα λέω ότι δεν έχουν την ευκαιρία να αποφεληθούν από τι εξελίξει. Ατενίζοντας λοιπόν το μέλλον, χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική για τι ανανεώσιμε, οι οποίες αυτές οι ίδιες αντιπροσωπεύουν το μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευθυνότερες και αυτό θα γίνουν και πιο δημοφιλείς πολύ σύντομα. Πρέπει όμως να τις προαγάγουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υποφύγουμε ζημιογόνους ανταγωνισμούς μεταξύ κρατών μελών στον τομέα. Ένα κατακλείδι θα λέγω ότι οι σημερινές συζητήσεις απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας είναι μια πολυσχηδής διαδικασία. Χαίρομαι προκειμένου που κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας έγιναν πολύ σημαντικά βήματα προς τα εμπρός στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων. Ελπίζω ότι και οι επόμενες Προεδρίες θα συμβάλλουν στην πορεία αυτή. Για άλλη μια φορά, παρακαλώ την Αντιπρόεδρο, την κυρία Τόγια, να μας πει δύο λόγια για τη συζήτηση. Ε. Ευχαριστώ. Να πω κάποια συμπερασματικά λόγια για την ολοκλήρωση αυτή τη ημερίδας. Μπορούσα να παρακολουθήσω ένα μόνο τμήμα, όμως με ενημέρωσαν ότι ήταν ιδιαίτερα έντονη η συζήτηση. Σήμερα το πρωί θα ήθελα κυρίω να ευχαριστήσω την Προεδρία της Λιθουανίας που είχε την ιδέα και πρότεινε και ανέλαβε και την πρωτοβουλία για αυτή την ε, κοινή συνεδρίαση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την εξαιρετική ιδέα και ευχαριστούμε και για την ε, συνεργασία μας ε, στα πλαίσια αυτής της Προεδρίας. Ολοκληρώσαμε μαζί σας πάρα πολύ σημαντικούς φακέλους που θα χαρακτηρίσουν την ευρωπαϊκή πολιτική της επόμενης επταετίας. Ήταν ιδιαίτερα λοιπόν καρποφόρος η συνεργασία όχι μόνο στο ενεργειακό τομέα αλλά και σε άλλα ζητήματα. Έτσι λοιπόν ε, χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτούς τους μήνες κοινή δουλειά ε, και ευχαριστώ και τον ε, συνάδελφο, τον κύριο Σαμαϊτάκης, γιατί προείδρευσε σήμερα και τον ευχαριστώ και για τις παρεμβάσεις του το πράτο αυτό εξ ονόματος ε, και όλων των συναδέλφων και της ε, κυρίας Σαρτόρη εν μέρη είδατε ε, ότι οι συνάδελφοι που ήταν εισηγητές ε, με πάθος ε, έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Αγοράς Ενέργειας και πρόκειται για ένα μεγάλο έργο αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια πιο καθαρή και πιο πράσινη οικονομία. Εγώ ελπίζω ότι η ευρωπαϊκή πολιτική θα εμπλουτίζεται όλο ένα και περισσότερο από αυτές τις ε, στιγμές ε, συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων, γιατί αυτό είναι το πνεύμα της συνθήκης της Λισαβόνα. Ε, και Πρόκειται για μια δουλειά που πρέπει να γίνεται από τα κοινοβούλια. Θέλουμε να δούμε τη συμμετοχή και κατά τη διάρκεια της λήψης αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για μας τους Ευρωπαίους γιατί πραγματικά συντονίζουμε τις απαιτήσει, τα προβλήματα και την εξέβρεση λύσεων. Ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες στα διάφορα κράτη-μέλη, είναι διαφορετικές οι συνθήκες, αλλά τελικά έχουμε την βαθιά αντίληψη ότι είναι ιδιαίτερα κοινά τα προβλήματα και ότι μόνο με μια κοινή πολιτική θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Αν και στον ενεργειακό τομέα το μείγμα των διάφορων λύσεων είναι εθνική επιλογή. Όμως για να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις εθνικές επιλογές φυσικά θα πρέπει να προχωρήσει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Κάτι δεύτερο, θα το πω πολύ σύντομα, το αναφέρατε κι εσείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εργαζόμαστε από κοινού για το θέμα της ενέργειας, γιατί χρειαζόμαστε την ενέργεια για να έχουμε και πιο αποτελεσματικές βιομηχανικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πολιτικές για την ανάπτυξη γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε ανάπτυξη ε, στην Ευρώπη ούτε εκ νέα εκβιομηχάνηση. Και οι περιβαλλοντικές πολιτικές ε, είναι ένα άχθος, είναι ένα στοιχείο εξισορρόπησης ή μπορούν να είναι ένα στοιχείο για εξέβρεση νέων ευκαιριών. Ακούσαμε τι συμβαίνει σήμερα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, ε, αναφερθήκατε στο ότι πρέπει να ενισχύσουμε την έρευνα για να έχουμε περισσότερη καθαρή ενέργεια. Θέλω να υπερθυμίσω σε όλους τους παρόντες ότι στο πρόγραμμα Ορίζοντας, Horizon, έχουμε του συναδέλφους που ήταν είτε σκιώδες είτε εισηγητές, στο πρόγραμμα ε, αυτό υπάρχει και ένα κεφάλαιο εντελώς καινούριο. Πώς ε, θα εξυπηρετήσει η έρευνα τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας ε, και το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και το ενεργειακό ζήτημα βρίσκονται στο επίκεντρο. Έτσι λοιπόν με το πρόγραμμα Horizon δίνει ήδη απαντήσεις η Ευρώπη υπό το προφίλ της αποδοτικότητας όλων των τομέων όπου θα εφαρμοστεί κατόπιν θα έχουμε και τη δράση των κρατών μελών, των ιδιωτικών και των δημοσίων φορέων, των κυβερνήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ακαδημαϊκών, των πανεπιστήμιων. Όλοι αυτοί θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά που θα τεθούν στη διάθεσή τους μέσω του προγράμματος. Ευχαριστώ σήμερα όλους τους συμμετέχοντες, τον ε, κύριο Μπλοκ, τον κύριο Μπέγκερ και ε, θα ήθελα να σας πω ότι οι διαφάνειες θα διατεθούν από τη γραμματεία σε όλους τους συμμετέχοντες. Και θα ήθελα να σας ευχηθώ και καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Πιστεύω ότι ήταν πολύ παραγωγική η ημέρα μας και δύσκολη. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους διερμηνείς σας ευχαριστούμε και εμείς. Και για να συνοψίσουμε, όσο χρόνο και να αφιερώνουμε στις συζητήσεις μας, όσο χρόνο και αν ε, δαπανούμε στις συζητήσεις για την ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ή την πυρηνική ενέργεια, την επόμενη εβδομάδα έχουμε Χριστούγεννα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να στολίσουμε το χριστουγεννιατικό δέντρο στο σπίτι μας. Επομένως θέλω να σας ευχηθώ. Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές ε, και να έχετε φως στη ζωή σας.